Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καθίστε παρακαλώ. Ε, εσείς που δεν παρακολουθήσατε που δεν παρακολουθήσατε το τμήμα και κλεισμένων των θυρών που μόλις ολοκληρώθηκε, καθίστε παρακαλώ. Call for your attention, please. Παρακαλώ την προσοχή σας. Προσέξτε παρακαλώ. Καθίστε στις θέσεις σας και να υπάρξει αρκετή ησυχία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο μετά από την κεκλεισμένο των θυρών τώρα στην ανοιχτή συνεδρίαση με το σημείο 10 την Ευρωπαϊκή Διάσταση στον Αθλητισμό και παρουσίαση ενός σχεδίου γνωμοδότησης από την κυρία Εμίν Μποσκούρτ όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση στα αθλήματα. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με την ίδια την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την διάσταση την ευρωπαϊκή στον αθλητισμό υπό το ευρύτερο πλαίσιο και με τις κοινωνικές επιπτώσεις και οικονομικές επιπτώσεις αλλά και κάποιες άλλες πτυχές που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες όπως ως Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Η κυρία Μποσκούτ έχει τον λόγο στη συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε. Η έκθεση αυτή το σχέδιο γνωμοδότησης ε, βασίζεται στο άρθρο 165 της ε, Συνθήκης Λισαβόνας που δημιουργεί κάποιες αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού και ο ρόλος της ε, Επιτροπής μας είναι πάρα πολύ σημαντικός εάν δούμε κάποια πράγματα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την διαφθορά στον αθλητισμό, την απάτη, παραδείγματος χάρη το στήσιμο αγώνων και το ξέπλυμα χρημάτων. Εάν διαβάζει κανείς την εφημερίδα βλέπουμε πως ε, το φαινόμενο αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και αλλού. Επίσης υπάρχει εμπόριο ανηλίκων ανθρώπων, υπάρχει εμπόριο ουσιών ντόπινγκ και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρξει και πολέμηση των διακρίσεων. Οπότε νομίζω πως είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Έχω προετοίμασα τις προτάσεις μου μετά από πολλές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, ε, Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, ε, ε, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επισκέφθηκα την UEFA και τη FIFA. Είχα συζητήσεις με την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τους λεγόμενους οργανισμούς του στοιχήματος. Οπότε είναι μία γνώμοδότηση, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει πως είναι περιορισμένη όσον αφορά το, το πλαίσιο και την έκταση, αλλά βλέπετε τις παρατηρήσεις που έχω κάνει στο κείμενο. Για τα υπόλοιπα σημεία, εγώ και ελπίζω και εσείς θα υποβάλω τροπολογίες. Ασχολήθηκα λοιπόν με την απάτη και το στήσιμο αγώνων αφενός και αφετέρου με το ντόπινγκ. Γιατί Βλέπετε πως είναι πάρα πολύ επίκαιρα αυτά τα θέματα και έχουν πάρα πολύ επιβλαβείς επιπτώσεις στον αθλητισμό. Αν δείτε το στήσιμο των αγώνων βλέπετε πως έχουμε και πρακτικές της μαφίας όπως το ξέπλυμα χρήματος, εμπόριο ανθρώπων και άλλες ε, δραστηριότητες που συνδέονται. Οπότε θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρξει εισαγωγή στο ποινικό δίκαιο όλων των κρατών μελών της έννοιας και του ορισμού, της απάτης, ε, του αθλητισμού και η Κομισιόν επίσης θα πρέπει να κάνει το ίδιο γιατί το στήσιμο αγώνων σε κάποια κράτη-μέλη τιμωρείται, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν ε, υφίσταται και άρα συχνά ξεφεύγουν ε, ατιμόρυτοι οι ένοχοι ή με έλαφρες ποινές. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβει την απάτη του αθλητισμού στην καταπολέμηση της διαφθοράς η Κομισιόν, την οποία συζητούσαμε σήμερα το πρωί. Οι δε οργανώσεις ε, του αθλητισμού συχνά κάνουν το εξής, δίνουν την οργάνωση σε κάποιους άλλους ε, υπομορφήν υπεργολαβίας. Εκεί πέρα δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος αυστηρός έλεγχος και άρα αν δείτε το τι γίνεται, έχουμε κάποιες σκιώδεις ε, οργανώσεις οι οποίες ε, έχουν την έδρα τους στην ε, Ταϊλάνδη, οι οποίες οργανώνουν και στείνουν αγώνες σε κράτη-μέλη περίεργα πράγματα. Υπήρχαν Ρώσοι πράκτορες μπλεγμένοι σε αυτές τις υποθέσεις, πράγματα τα οποία πρέπει να σταματήσουν. Επιπλέον θα πρέπει οι φορείς του αθλητισμού να συνεργαστούν περισσότερο με την Europol και τέλος η Europol θα πρέπει να συνεργαστεί με κοινέ ομάδες έρευνας για να ερευνήσει επαρκώς το θέμα αυτό το οποίο υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, κάτι το οποίο συνέβη στην Φινλανδία. Εκεί πέρα συνελήφθησαν άνθρωποι ε, ενός ασιατικού συνδικάτου του εγκλήματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε δραστηριότητα σε πάρα πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες και η Eurojust θα πρέπει να δει μετά την ε, δικαστική πτυχή. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των φορέων του αθλητισμού και των εταιριών του στοιχήματος για να ξεκαθαρίσει ο κλάδος από τις ε, βλαβερές επιπτώσεις του συστήματος για να παραμείνει καθαρέως ο όλος κλάδος και να υπάρχει και η αίσθηση εμπιστοσύνη του κοινού πως ε, δεν υπάρχει απάτη. Αυτό το οποίο λοιπόν δεν υπάρχει στην ε, έκθεση είναι πως δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτό, αλλά σημαντικά θέματα είναι τα αστικά δικαιώματα των αθλητών, εμπόριο ανηλίκων αθλητών και οι διακρίσεις. Επίσης το ντόπινγκ είναι κάτι το οποίο θέλω να τονίσω. Είναι σημαντικό να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ χωρίς να παραβιάσουμε τα δικαιώματα στην ε, ιδιωτική ζωή και τα υπόλοιπα ατομικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Οπότε θα πρέπει να ορίσουμε ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Δεύτερον, οι μάνατζερ των παιχτών οι οποίοι ασχολούνται με ανήλικους παίχτες. Σε ένα μόνο έτος, το 2010, είχαμε 1.100 ανηλίκους οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο συμβολέων. Είχαμε κάποιες συμφωνίες λοιπόν και φαίνεται πως ε, θα πρέπει να περιοριστεί το εμπόριο ανηλίκων ε, παιχτών και να λαμβάνει χώρα μόνο κατ' εξαίρεση. Όταν μιλάμε λοιπόν για 1100 άτομα δεν μιλάμε πλέον για εξαίρεση. Και αυτό πρέπει να, ανασταματήσει λοιπόν να περιοριστεί σε ένα μίνιμουμ και να το δούμε κατά περίπτωση αυτή τη στιγμή μπορεί ο καθένα να γίνει μάνατζερ παιχτών χωρίς κάποια εκπαίδευση. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να υπάρξει ε, κάποια εγγραφή σε ένα αρχείο και κάποια επαγγελματικά προσόντα. Τέλος, διακρίσεις θα πρέπει να οριστούν κάποιες βέλτιστες πρακτικές από την Κομισιόν για την καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά στην ανακοίνωση τη σχετική βλέπετε πως δεν υπάρχουν κάποιες δράσεις για να υποστηριχθούν όλα αυτά. Οπότε το ερώτημα είναι τι θα κάνει στην πράξη η Κομισιόν για να καταπολεμήσει το μίσος, το ρατσισμό και όλα αυτά στα γήπεδα. Οπότε νομίζω πως ε, έχουμε εδώ πέρα τη βάση για να καταλήξουμε σε μια αρκετά καλή ε, γνώμοδότηση. Σας ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ τώρα. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει το θέμα, μπορεί να συζητήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Κάποιος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, παίρνω το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτριά μας και να συμφωνήσω με όλα όσα ανέφερε και να ενώσω και εγώ τη δική μου φωνή στα όσα είπε για τα θέματα της απάτης και της διαφθοράς στον αθλητισμό. Τους περασμένους μήνες στην Ελλάδα αντιμετωπίσαμε ε, μια αντίστοιχη ε, πολύ σημαντική υπόθεση. Ε, προέκυψε ότι παράγοντες ομάδων δημιουργούσαν τις ε, προϋποθέσεις για να στείνουν αγώνες, να προδιαγράφουν αποτελέσματα, ε, στοιχήματα πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες, ε, αυτό που αναφέρατε και προηγουμένως. Το περίεργο δε ήταν, και είναι γιατί η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και έχει επιληφθεί και η δικαιοσύνη, ότι οι ίδιοι παράγοντες ήταν ιδιαίτερα δικτυωμένοι και στην εθνική ομοσπονδία για το ποδόσφαιρο και στην διοίκηση του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο. Την περίοδο λοιπόν εκείνη και μέχρι σήμερα πολλοί ήταν εκείνοι ε, που ανέφεραν ότι είναι ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν εντονότερες πρωτοβουλίες και να υπάρξουν ε, πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της εποπτείας και του ελέγχου ε, τέτοιων περιστατικών και της λειτουργίας των ομοσπονδιών και ευρύτερα των εθνικών δομών για τα αθλήματα και πράγματι η έκθεση αυτή της Επιτροπής Παιδείας που και εμείς νομοδοτούμε έρχεται σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο ε, σε ένα σημείο που έχουμε αρμοδιότητα βάσει θήκης Λισαβόνας και σε ένα σημείο που και οι ίδιοι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Πιστεύω πως ε, θα πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών και αυτή η ημερομηνία είναι Δευτέρα Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18.00. Συμφωνείτε με την προθεσμία αυτή. Ωραία. Προχωράμε. Περνάμε στο σημείο υπαρθμών 11 Πρόκειται για τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σέγγεν και τη σύμβαση ε, εφαρμογή τη συμφωνία του Σέγγεν. Κοιτάξτε, η συγγητή ε, είναι ο συνέλφος κ. Παπα-Νικολάου και το ιστορικό έχει εξή. Πριν από μερικού μήνε η Κομισιόν ανέκρινε μια πρόταση για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σέγγεν και τη σύμβαση εφαρμογή τη Συμφωνία Σέγγεν. Θα ακούσουμε αυτή την ε, παρουσίαση, η οποία ήταν ιδιαίτερα επίμαχη ευθύ εξ αρχή. Θα ακούσουμε λοιπόν την Κομισιόν και μετά θα ακούσουμε τον συγητή μα, ε, κύριο Πανικολάου, την Πολωνική Προεδρία και θα ακολουθήσουν τα μέλη. Αλλά φαίνεται πως ε, βρισκόμαστε σε αναμονή του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα, κατά 10 λεπτά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, να διακόψουμε για ένα δεκάλεπτο, συμφωνείτε, προκειμένου να αφηχθεί και η Κομισιόν. Λοιπόν, σωστό θα ήταν λοιπόν, μια που Θα πρέπει να ακούσουμε την Κομισιόν πρώτα. 10 λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ. Ξέρουμε πως κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αλλά καμιά φορά μπορεί και να είμαστε μπροστά από το πρόγραμμα. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μία ετοιμότητα να παρέμβει κανεί. Εν πάση περιπτώσει καλωσορίζουμε την Κομισιόν που είναι σημαντική για την παρουσίαση της πρότασης τροποποίησης του κώδικα Σέγγεν και της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σέγγεν. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την Κομισιόν και μετά τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον εισηγητή μας, για να ξεκινήσει η συζήτηση η κυρία Μόνικα Μοσόμερα, από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη. Συνήθως έρχομαι νωρίτερα, αυτή τη φορά δεν, δεν μπόρεσα. Θα είμαι σύντομη και ακριβής ε, με την παρουσίαση των αλλαγών του κώδικα συνόρων Σέγγεν και της σύμβασης ε, Σέγγεν όπως υιοθετήθηκαν αυτές οι αλλαγές από την Κομισιόν τον Μάρτιο. Να υπογραμμίσω πως ε, Πρόκειται για μια τροποποίηση που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο και δεν αποτελεί απάντηση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στην Ολομέλεια δήλωσε πως θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις τον Σεπτέμβριο οπωσδήποτε, αλλά δεν πρόκειται για την τροποποίηση αυτή μετά το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να επανέλθω λοιπόν στην ουσία της πρότασης του Μαρτίου. Γιατί γίνεται αυτή η πρόταση. Πρόκειται για μία αναθεώρηση του κώδικα συνόρων Σέγγεν μετά από πέντε έτη πρακτικής εφαρμογής. Για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να δούμε τι μας λένε οι άνθρωποι που το εφαρμόζουν, τι λειτουργεί σωστά, ποιες είναι οι βελτιώσεις που χρειάζονται. Επίσης η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να, επίσης να απαντήσει αφενός και για τις φραγίδες αυτέρου για την επανεισαγωγή συνοριακών ελέγχων. Θα δείτε τα συμπεράσματα και τις πρακτικές εμπειρίες που έχουν μεταφραστεί στην τροποποίηση αυτή. Όπως είπα λοιπόν δεν πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία, οπότε οποιαδήποτε ιδέα συστήματος εισόδου-εξόδου ή οτιδήποτε άλλο μετά από την παρακίνηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν συμπεριλαμβάνεται. Πρόκειται εδώ με τεχνική τροποποίηση. Επίσης δεν πρόκειται για κωδικοποίηση ή αναδιατύπωση για την οποία επιφυλασσόμεθα. Το σκεπτικό εδώ πέρα της τροποποίησης είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολύνουμε περαιτέρω τα πράγματα για να μην δημιουργούμε εμπόδια για το να διασχίζει κανείς τα εξωτερικά σύνορα. Οι βασικές αλλαγές αφορούν οι οριζόντιες. Είναι η προσαρμογή στην συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε τώρα πλέον γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης ε, αλλάξαμε τις παλαιές διατάξεις στο νέο καθεστώς ε, της ε, συνθήκης Λισαβόνας. Έχουμε λοιπόν όπως συμφωνήσαμε μια διατύπωση για τις πράξεις κάτω εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ μέσα. Θα βρείτε λοιπόν την τυποποιημένη διατύπωση για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση και τρίτη οριζόντια αλλαγή είναι ευθυγράμμιση με την λυπή κοινοτική νομοθεσία που έχει εντωμεταξύ οθετηθεί δηλαδή το τον κώδικα θεωρήσεων ε, και την οδηγία επιστροφής. Θα δείτε λοιπόν αυτή την ευθυγράμμιση στο άρθρο 5 του κώδικα συνόρων Σέγγεν όπου μιλάμε για τα ταξιδιωτικά έγγραφα και στο άρθρο 11 όπου μιλάμε για την παραμονή ε, ατόμου εκεί που γίνεται λόγος για την οδηγία επιστροφής και έχουμε επίσης ενημερώσει τις αναφορές που υπάρχουν στον, κανόνα, στον κανονισμό περιστατιστικής. Αυτά για να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινοτική νομοθεσία στον μεταξύ. Επί της ουσίας, μπορώ να τονίσω μόνο τα σημαντικότερα, θέλαμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία, γι' αυτό συμπεριλάβαμε και τις ε, αποστολές εμπορευμάτων στο καθεστώς των εσωτερικών συνόρων, οπότε να μην υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους στο μέλλον. Επιπλέον, κάποιες κατηγορίες ατόμων, ε, όπως παραδείγματο χάρη το προσωπικό των σιδηροδρόμων δεν ανάγκη να σφραγίζονται κάθε φορά τα διαβατήριά τους, κάθε φορά περνάνε τα σύνορα. Επίσης, σκεφτήκαμε πως θα είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι υποχρέωση, να έχουμε διαφορετικές ουρές στα τελωνιακά φυλάκια για να μην υπάρχει πρόβλημα σε όσους περνάνε χωρίς βίζα. Επίσης εκπαίδευση των σύνοριοφυλάκων για να ανοιχνεύουν ευπαθείς ομάδες όπως άτομα τα οποία είναι θύματα σώματεμπορίας να ευαισθητοποιήσουμε λοιπόν τους συνοριοφύλακες σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και τέλος η Κομισιόν θεωρεί πως μπορεί να καταργηθεί η υποχρέωση αναφοράς καθώς δεν χρησιμοποιείται πολύ από τα κράτη-μέλη. Σημαντικό επίσης είναι η δημιουργία κανόνων για κοινά συνοριακά φυλάκια μεταξύ κρατών μελών και τρίτης χώρας. Η δυνατότητα αυτή δεν ε, προβλεπόταν ρητός στον κώδικα συνόρων Σέγγεν, οπότε έπρεπε να εισαχθεί για να δημιουργηθούν συνέργειες εδώ πέρα. Να τονίσω εδώ πέρα πως δεν είναι θέμα του να αναλάβει τις ε, πύλες ε, εισόδου και εξόδου μιας τρίτης χώρας σε ένα κράτος μέλος ή αλλά είναι το να υπάρχει μία υποδομή στη μία πλευρά των συνόρων και να μην σταματάνε δύο φορές ε, οι άνθρωποι π.χ. και στην πλευρά της Πολωνίας και στην πλευρά της Ουκρανίας. Αλλά για να καταστεί αυτό δυνατόν χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες και ιδιαίτερα όσον αφορά το να εγγυηθούμε την πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου ειδικά όταν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι σε επικράτεια τρίτους, τρίτου κράτους ε, ή όταν ε, ε, κάνει συνοριακούς ελέγχους το τρίτο κράτος στην επικράτεια ενός κράτους μέλους. Αυτά και αναμένω την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή για την παρουσίαση, την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την εισαγωγή και την παρουσίαση που μας έκανε. Να προσθέσω στα όσα είπε τα εξής. Ε, έχουμε ενώπιον μας μία πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία ε, έρχεται να επικαιροποιήσει τον κανονισμό που διέπει ε, το Σέγγεν από το 2006. Πέντε χρόνια μετά λοιπόν, ε, με βάση και, τα, και, τις νομο, και τις νομικές αλλαγές, τις αλλαγές σε νομικό επίπεδο που είχαμε, ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως υπόθηκε, με τον κώδικα θεωρήσεων του 2009, με τις αξιολογήσεις από την πρακτική εφαρμογή, με τις διατάξεις για τις φράγκες των ταξιδιωτικών εγγράφων και διάφορα άλλα όπως αναφέρονται, ε, καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε και να εναρμονίσουμε αυτά τα κείμενα ε, προκειμένου να μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις προκλήσεις. Αυτό βεβαίως που πρέπει να διευκρινίσουμε στην πρώτη συζήτησή μας είναι ότι αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2009 ε, λίγο πριν ε, λάβουν χώρα όλες οι εξελίξεις που παρακολουθούμε όλοι μας τους τελευταίους μήνες. Την αναφορά δηλαδή που γίνεται στο Σέγγεν μετά τις μεγάλες ροές που είχαμε από τη Βόρειο Αφρική στην Ιταλία και τη μετακίνησή του στη Γαλλία, την στάση τότε που είχαμε ε, από τις χώρες αυτές, στη συνέχεια την ε, τοποθέτηση της Δανίας και την επαναφορά συνοριακών ελέγχων, η τοποθέτηση μετά του Συμβουλίου του Ιουνίου και η πρόσκληση που έκανε, όπως αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, στην στην πρωτοβουλία που αναμένουμε για την ε, δυνατότητα επαναφοράς συνοριακών ελέγχων και εν ολίγης τους τελευταίους μήνες ε, ξεκίνησε ξανά μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο μας για το κεκτημένο Σέγγεν, μια βασική αρχή που διέπει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κεκτημένο το οποίο βεβαίως όλοι από την πρώτη στιγμή ε, υποστηρίζουμε και τοποθετηθήκαμε καθαρά το κοινοβούλιο μας με όλα του τα κείμενα και όλες τις τοποθετήσεις ε, σε σχέση με τη διαφύλαξη του κεκτημένου αυτού αλλά και βεβαίως τη διεύρυνση του χώρου Σέγγεν με την ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έχουμε αποφασίσει στο κοινοβούλιο μας αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη την ανταπόκριση του Συμβουλίου παρότι από ό,τι προκύπτει από όλες τις αναλύσεις πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή του στο χώρο Σέγγεν. Ε, επομένως, ε, πέραν της τεχνικής επεξεργασίας που έχουμε να κάνουμε στο ε, κείμενο αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλο αυτό το περιβάλλον. Οι πολίτες αναμένουν από εμάς καθαρές απαντήσεις στα θέματα αυτά ε, και να διευκρινίσω και εγώ τούτο, ότι σε μια τέτοια έκθεση βεβαίως όταν αναφέρουμε και ξεκινάμε την παραδοχή ότι οι περισσότερε αλλαγέ είναι τεχνικού χαρακτήρα, αυτό ενδεχομένως διευκολύνει στο να μπορέσουμε να έχουμε ε, συμφωνία, να έχουμε ομοφωνία και συνένεση μεταξύ μας και να μην υπάρχουν ενδεχομένω σημαντικέ πολιτικέ διαφοροποιήσει. Όμως, οφείλουμε ως Κοινοβούλιο να καταθέσουμε και την αγωνία μας αυτή και παρακαλώ την Επιτροπή αλλά και την Προεδρία αν έχουν κάτι περισσότερο να μας πούν τόσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχουν για τη νέα τροποποίηση του κώδικα ε, σε σχέση με την ε, ανακοίνωση του Συμβουλίου του Καλοκαιριού αλλά και την άλλη τροποποίηση που αναμένουμε και εκείνη ε, που δεν έχει σχέση βεβαίως με αυτή την έκθεση ε, για το ζήτημα του της έξυπνης διαχείρισης των συνόρων όπως λέμε, αυτό θα ήταν σημαντικό προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα και να μπορέσουμε να κατευθύνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ε, τη δράση μας και τις δικές μας διαδικασίες. Ε, βεβαίως δεν διαφωνεί κανείς ότι με αυτήν την ανακοίνωση επιδίωξη είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, είναι η διευκόλυση των διαδικασιών, ε, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα. Σε αξιολογήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα έχουν υπάρξει σημαντικές διαπιστώσεις και εμείς στο κοινοβούλιο μας συζητήσαμε διεξοδικά το προηγούμενο διάστημα τα θέματα αυτά με τον εξαιρετικό συνάδελφο που είναι και ο, πλέον ειδικό στα θέματα Σέγγεν, τον κύριο Κοέλη, ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ε, και ε, αποφεύγω και εγώ να πω περισσότερα σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα. Νομίζω τα περισσότερα τα ανέφερε η ε, εξαίρετη εκπρόσωπος της Επιτροπής να ε, προσθέσω μόνο ε, το εξής. Σε ό,τι αφορά την, και να το εξηγήσω αυτό συναδέλφους και να κλείσω έτσι την πρώτη μου εισαγωγή σε αυτό και παρακαλώ για την όποια δική τους για τον όποιο δικό του σχολιασμό στα θέματα αυτά. Στην πρόταση τροποποίησης έχουμε δύο βασικά άρθρα η, πρώτη αφορά τις αλλαγές στον κώδικα των συνόρων, στον κώδικα Σέγγεν και η δεύτερη αναφέρεται στην διαγραφή δύο άρθρων και μιας παραγράφου, εν πάση περιπτώσει στις αλλαγές που, ε, ε προκύπτουν στην σύμβαση της εφαρμογής της συμφωνίας του Σέγγεν. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατευθύνσεις οι οποίες έχουμε στις αλλαγές ε, που καλούμαστε να κάνουμε. Ε, προφανώς πρέπει να ενημερώσουμε και την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι η δική μας πρόθεση είναι το ε, κεκτημένο Σέγγεν να ε, διατηρηθεί στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Η επιδίωξή μας είναι βεβαίως να μην υπάρχει γραφειοκρατία, βεβαίως να διευκολύνουμε όσο γίνεται τις διαδικασίες και τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο να κινούνται ανεμπόδιστα εντός της Ένωσης. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε ισχυρά και ασφαλή εξωτερικά σύνορα, ε, διαδικασίες τέτοιες που να διασφαλίζουν ότι ακριβώς επειδή η αλληλεγγύη και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ μας είναι τέτοιες και με τεχνικούς αλλά και με πολιτικούς όρους ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ε, το εσωτερικό της Ένωσης είναι ασφαλές και δεν υπάρχει λόγος για ανασφάλειες και για προβληματισμούς όπως αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες. Δεν προχωρώ περαιτέρω κύριε Πρόεδρε σε αυτήν την φάση. Αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις εισαγωγικέ παρατηρήσει και των συναδέλφων και βεβαίως και εγώ ε, δεσμεύομαι και ενώπιον σας και ενώπιον του Συμβουλίου και της Επιτροπή να καταθέσω τον καλύτερο με αυτό για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ. Thank you. Now maybe we could hear... Τώρα ίσω θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι από πλευρά τη πολωνική Προεδρίας εκπροσωπείται από τον κύριο Μιλόσλαβ Νούτσικ. Ίσως θα θέλετε να μας πείτε εσείς ε, κάποια πράγματα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μιλόσλαβ Νουτσίκ είναι το όνομά μου. Σύμβουλος και εκπρόσωπος ε, της ε, Πολωνίας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιος για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αρμοδιότητα αυτή οι τροπολογίες για τον κώδικα Σέγγεν ανήκουν στην δική μου αρμοδιότητα. Για το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις απόψεις της, για τις τροπολογίες στον κώδικα Σέγγεν και στη σύμβαση για την τη ζώνη Σέγγεν και διεξήχθη μια γενική συζήτηση. Μετά από αυτή τη συζήτηση είχαμε τα εξή συμπεράσματα. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν ως προς την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κώδικας Σέγγεν τον Ιούλιο 2011 μια πρώτη συνεδρίαση, πρώτη συνάντηση μια ειδική ομάδα για συνοριακού ελέγχου διεξήχθη υπό την Πολωνική Προεδρία και η πρώτη ανάγνωση του κειμένου έγινε. Σε πέντε συνεδριάσει που έγιναν, που προγραμματίστηκαν αυτή τη ομάδα, η επόμενη θα γίνει στι 15 Σεπτεμβρίου και οι επόμενες συνεδριάσεις 13 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο κατά τα τέλη τη Πολωνική Προεδρία, θα υποβάλουμε έκθεση ω Πολωνική Προεδρία για το έργο αυτή τη ομάδα εργασία και για τις τροποποιήσεις στον κώδικα Σέγγεν και τη σύμβαση για το Σέγγεν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι η Πολωνική Προεδρία θα δράσει με κάθε δραστήριο τρόπο επί αυτού του σημαντικού ρυθμιστικού έργου και θα σας διασφαλίσω ότι θα είμαστε πάντα σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε τακτά διαστήματα θα έχουμε συναντήσεις με τον εισηγητή, τον κύριο και στη συνέχεια ο κοινό μας στόχος ποιος είναι. Ο κοινό μας στόχος είναι να επιτύχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο είναι εφικτό να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Και τώρα κάποια χέρια έχουν εγερθεί. Ξεκινάμε με την κυρία Μποσκούρτ. Έχετε τον λόγο πρώτη κυρία Μποσκούρτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστήσω και τον ε, κύριο παπα για την παρουσίαση αυτή έχω κάποιες ε, ερωτήσεις για την πρόταση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ερωτήσεις για το 1.2.1 και 1.2.2 τα σημεία αυτά. Εκεί πέρα αναφέρεται πως ε, για πρακτικούς ε, λόγους ε, στις περιπτώσεις στις οποίες γίνονται έλεγχοι μπορεί αυτοί να παραληφθούν. Γιατί το προτείνει αυτό η Κομισιόν, ποιοι είναι αυτοί οι πρακτικοί λόγοι τους οποίους αναφέρει και το ερώτημα είναι τι θα γίνει εδώ πέρα, θα αυξηθούν οι έλεγχοι ή όχι. Επιπλέον, αναφέρεται πως ε, κατά παρέκκληση των άρθρων 4 και 7 ε, δεν θα γίνεται έλεγχος σε άτομα τα οποία επιβαίνουν σε πλοία χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι συνοριοφύλακες ε, δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο του πλοίου και των επιδενόντων ε, για κινδύνους εσωτερικής ασφάλειας και παράνομης μετανάστευσης. Αυτό τι σημαίνει θα ισχύσει το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών σε αυτή την περίπτωση. Επίσης η πρόταση περί εκπαίδευσης ε, είναι σωστή, αλλά αυτό σημαίνει πως θα περιοριστεί μόνο σε ανηλίκους ε, και τέτοιες ομάδες. Τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι χρήζουν ε, διεθνούς προστασίες Και για να αναφερθώ και σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου, μιλάμε για αλλαγή του κώδικα συνόρων του 2006, αλλά εδώ πέρα μιλάμε και για την Συμφωνία Σέγγεν, αναφέρεται μάλλον και η Συμφωνία Σέγγεν. Τι εννοεί ακριβώς εδώ πέρα η Κομισιόν σε ποιο πλαίσιο πρέπει να δούμε αυτή την ε, αλλαγή σε σχέση με τις ε, υπόλοιπες προτάσεις ε, αλλαγής της συνθήκης έγκεν που συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος, για τις διμερείς συμφωνίες για τις οποίες κάτι είπε η Κομισιόν για το πώς θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, αλλά το ερώτημά μου είναι πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο στην πράξη, γιατί μου ακούγεται εξαιρετικά περίπλοκο πώς θα γίνουν ακριβώς τα πράγματα. Αυτά θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριο Σκέκοπ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω κάνα δύο πράγματα για το, τη θεμελιώδη φύση του έργου εδώ πέρα της Κομισιόν. Γιατί σαφώς, όπως υπόθηκε από την αρχή, δεν μιλάμε για την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε το 2006. Οπωσδήποτε δεν είναι ίδια η Ευρώπη. Είχαμε την συνθήκη της Λισαβόνας, τα επιπλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλαγές στη μετανάστευση, αλλαγές ε, στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, τις πιέσεις από την Βόρεια Αφρική κτλ. λοιπά Οπότε η πρόταση της Κομισιόν εμένα μου φαίνεται κάπως άτολμη. Βεβαίω κάποιοι θα μου πούν ε, να κοιτάτε τη δουλειά σα, κύριε Κέρκοπ γιατί ούτω ή άλλω το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Σέγγεν. Ήμουν υπουργό Συνόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευχαρίστω ε, να σα δώσω κάποιε συμβουλέ, Ίσως ενδιαφέρουν εσά περισσότερο από την ε, προηγούμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου, αλλά είναι σημαντικό και για το Ηνωμένο Βασίλειο να λειτουργεί σωστά η Σέγγεν και να έχουμε ευρωπαϊκά σύνορα. Εξίσου σημαντικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οπότε αυτό το οποίο έχω να πω έτσι γρήγορα κύριε Πρόεδρε είναι το εξή. Οπωσδήποτε αυτό αφορά κάποια ίσονο σημασία ζητήματα, ευθυγραμμισμού ορισμών ε, και κάποια άλλα πράγματα, αλλά περιλαμβάνει και απαιτήσει ε, παράλογε. δηλαδή να αναφέρονται νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που μπαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη. Πώς θα γίνει αυτό με ανοιχτά σύνορα γιατί τα πραγματικά ζητήματα υπάρχουν. Τα πραγματικά ζητήματα είναι η ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης της ε, Σέγγεν. Όπως ακριβώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει τα των συνόρων του για να αξιολογήσει τις νέες σύγχρονες απειλές. Θέλουμε ε, Σοβάρε μεταρρυθμίσει εάν είναι να ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα η Σέγγεν. Επίση υπάρχουν νομικές και τεχνικέ αλλαγές οι οποίες θα απαιτήσουν την ριζική αναθεώρηση από κάτω προς τα πάνω της Σέγγεν όπως τα ζητήματα εναρμόνισης βίζας, τα ηλεκτρονικά σύνορα, το σύστημα εισόδου-εξόδου στην Ένωση, το πρόγραμμα καταγεγραμμένων ταξιδιωτών της Ένωσης, επίσης ζητήματα όπως η συμφωνία η μου για τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών στο οποίο είμαι εισηγητή. Ε, κατόπιν πρέπει να δούμε την επανεισαγωγή συνοριακών ελόγχων από κάποια καρτιμέλη. Δεν αρκεί να ασκούμε κριτική στους Γάλλους ή Ιταλούς γείτονέ μας. Έθιξαν κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ πολλούς Ευρωπαίους και δεν έχει νόημα να λέμε ε, πως θα πρέπει απλά να ακολουθούν τη Σέγγεν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αντικατοπτρίσουμε αυτές τις αλλαγές, τις δυσκολίες και από τη βασική δομή της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων να δούμε τις προκλήσεις και να αναθεωρήσουμε ριζικά την Σέγγεν για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Αν αυτό είναι διατεθειμένη να κάνει η Κομισιόν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που έχουν ανησυχίες και με τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Σέγγεν όπως η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε εγώ θα σας ε, στηρίξω και αυτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι αρνητικοί για τη Σέγγεν και λένε όλα αυτά είναι μπουρδες και ευτυχώς που έχουμε δικά μας σύνορα, νομίζω πως είναι αφελής, γιατί όλοι ε, έχουμε την ανάγκη να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης και να αναπτύξουμε τις δημοκρατίες ε, στην Ευρώπη με τρόπο που θα μας ωφελεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νεντέλτσεβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο για την παρουσίαση για τα θέματα της μελλοντικής αυτής έκθεσης. Πιστεύω ότι ένας κανονισμός θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός στην ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων και μια διευκόλυνση για τους πολίτες να μπορούν να διασχίζουν, να περνούν τα σύνορα αυτά. Βρίσκω πολλές θετικές πτυχές στις προτάσεις αυτές όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο έκθεσης. Ακούσαμε πολλές λεπτομέρειες για τεχνικά θέματα, ειδικού όρους και προϋποθέσεις για διασώστες ομάδες διάσωσης που διασχίζουν τα σύνορα. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία. Η κοινή εκπαίδευση, κατάρτιση των σύνοριοφυλάκων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή την έκθεση, σε αυτή την πρόταση. Θα ζητούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο εξειδικευμένα να μας δώσει λεπτομέρειες όσον αφορά το σκέλος της κατάρτισης και εκπαίδευσης αυτών των συνοριοφυλάκων. Ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανηλίκων και θέματα ε, ατόμων που είναι θύματα εμπορίου ανθρώπων. Επίσης η ασυνόδευτη ανήλικη είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα και όλο και περισσότερη σημασία αποκτά, όλο και σπουδαιότερο γίνεται ως θέμα για την διαχείριση συνόρων. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πρόκληση. Είναι η μετανάστευση παιδιών, η διακίνησή τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, ε, σε άλλο εκτίθενται σε κινδύνους εκμετάλλευσης, κατάχρησης, κακοποίησης ακόμα αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν κίνδυνοι λοιπόν. Τι γίνεται σε σχέση με την κατάρτιση και εκπαίδευση. Καλύπτονται αυτές οι πτυχές όσον αφορά την εκμετάλλευση παιδιών για παράδειγμα και πολιτών εξάλλου εξίσου θα ήθελα να συστήσω, να επενέσω τις θετικές αυτές προτάσεις που βρίσκονται στην έκθεση του κυρίου Κουέλιο. Και εν τέλει υποστηρίζω την θέση που έχει υιοθετήσει ο κύριος Παπα-Νικολάου όσον αφορά τις τεχνικές προσαρμογές θεμάτων που δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Να τονίσω και να πω ότι φυσικά συμφωνούμε ότι αυτές οι τεχνικές προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν μέσα στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτό. Σε σχέση με το πρόβλημα, δεν αναφέρθηκε από πλευράς εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα της συμπερίληψης της ένταξης θεμάτων νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αυτό το πλαίσιο. Δεν άκουσα τίποτα σχετικά. Θα ήθελα να ακούσω κάποια σχόλια επ' αυτού του θέματος για την νομολογία του ΔΕΚ, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε σχέση και με την υποχρέωση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Όταν έχουμε πολίτες που ταξιδεύουν από ένα κράτος μέλος σε άλλος, σε άλλο. Θα ήθελα να ακούσω από το Συμβούλιο ποια είναι η αντίδρασή του σε αυτή την πρόταση. Είμαι υπέρ της κατάργησης σε σχέση με την υποχρεωτική αναφορά καταχώρηση όλων αυτών. Θα ήθελα να ακούσουμε όμως ποια είναι η θέση των άλλων ε, θεσμικών οργάνων. Επίσης έχω μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα ήθελα ακόμα να μου πείτε, κύριε, αν υπάρχουν κάποιες προθέσεις ε, να συζητηθούν οι αλλαγές στις ε, διεργασίες, στις διαδικασίες για τις, ε, την προσωρινή εισαγωγή συνοριακών ελέγχων ή όχι σε σχέση με τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Είμαστε λοιπόν αδειμονούμε να ακούσουμε από αυτού θέματα το δικό σας σχολιασμό. Ευχαριστώ. Από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μόσχαμερ, θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτά τα ερωτήματα. Η εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Όπως προσπάθησα να επεξηγήσω προηγούμενα, Αυτές οι τροποποιήσεις είναι ουσιαστικά τεχνικού χαρακτήρα. Υπήρξαν και συζητήσεις φυσικά για την περαιτέρω ανάγκη να ενισχυθεί, να τονωθεί ο χώρος Σέγγεν και στην ανακοίνωση της 4ης Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήχθη στη συνέχεια και συζήτηση στην Ολομέλεια του Ιουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον κύριο Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς για πιθανές τροποποιήσεις και σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για την ενίσχυση του χώρου Σέγγεν και του αντίστοιχου μηχανισμού. Θα απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτό λοιπόν θα τεθεί επί στο τραπέζι σας στο άμεσο μέλλον. Ακόμα δεν είναι αντικείμενο σε σχέση με την τροποποίηση που είχε εισαχθεί μετά τον ε, Μάρτιο. Και έτσι λοιπόν τα όσα συνέβησαν μετά έχουν αλλάξει το πλαίσιο. Αυτό όμω είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο είχε υιοθετηθεί το Μάρτιο. Και όσον αφορά τα ευφυή σύνορα, θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά με διαφορετικό τρόπο θα επανέλθει η Επιτροπή τον Οκτώβριο και θα σας ενημερώσει για τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις και ερωτήσεις για την τρέχουσα πρόταση Ελπίζω ε, να τις ε, έχω όλες ε, αυτές και να απαντήσω σε όλες και αν δεν απαντήσω διμερώς μπορούν να αποσαφινιστούν κάποια θέματα. Τώρα, για την αλλαγή των διαδρομών των, ουρο, της, διά, της ε, διάσχεσης ε, συνόρων ε, κάθε φορά που γίνεται αυτό μπορούμε ήδη σε ένα σταθμό σιδηροδρομικό μιας τρίτης άλλης χώρας να καλύπτονται οι ανάγκες. Τώρα για την κατάρτιση και εκπαίδευση φυσικά η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σημαντική Θέλαμε όμως να θέσουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι θα πρέπει οι συνοριοφύλακες να μπορούν να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν ευάλωτες ομάδες. Φυσικά όλα τα άτομα που χρήζουν αρρωγής και βοήθειας και γι' αυτό από πλευράς Frontex που διοργανώνει τέτοιου είδους μαθήματα για την κατάρτιση και εκπαίδευση στόχος μας ήταν να ενταχθεί ένα τέτοιο μάθημα και να υπογραμμιστεί η σημασία της ε, επαρκούς κατάρτισης και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε τα αντίστοιχα προγράμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, για τα θέματα που αφορούν το άρθρο 32 και το άρθρο 33 όσον αφορά επιτροπολογία. Είχαμε επιτροπολογία που προβλεπόταν ε, υπό διαδικασία που έχει αντικατασταθεί τώρα μέσω των κατεντολήν κατεξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με το άρθρο 32 και 33 η αναφορά στις κατεξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η διατύπωση που είχε συμφωνηθεί σε σχέση με τις διοργανικές συμφωνίες. Α, τέλος, αλλά σημαντικό, πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες για τις, ε, την κοινή διάσκηση συνόρων θα σέβονται τον κώδικα. Όσον αφορά τον συνοριακό κώδικα, τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού συναυθούν ολοκλήρωσα. Ελπίζω ότι κατάφερα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Αν εκκρεμούν κάποιες διμερώς είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ. Thank Now the Polish Mr. Σας ευχαριστώ. Τώρα η Πολωνική Προεδρία. Εσείς κύριε, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση ε, τέθη από φράσεις κυρία Στανόκα προς την Προεδρία. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Να σας ενημερώσω πως η Πολωνική Προεδρία θα εστιαστεί στο αίτημα της ε, Κομισιόν και θα εργαστούμε σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τώρα όσον αφορά την επανεισαγωγή των ε, εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα. Κοιτάξτε, αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον ε, κώδικα Σέγγεν σήμερα και μέχρι να υποβληθεί νέο αίτημα δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Ευχαριστώ από τον εισηγητή μας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους εκπροσώπους και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ε, νομίζω γίνεται αντιληπτό ότι όλοι κατατείνουμε στο ίδιο τελικό συμπέρασμα ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το χώρο Σέγγεν, να διαφυλάξουμε το κεκτημένο Σέγγεν να σταματήσουμε κάθε συζήτηση περί αμφισβήτησής του και ως εκ τούτου εφόσον και μέσα από αυτή την ε, τροποποίηση που επαναλαμβάνω έρχεται να εναρμονίσει ε, τα κείμενα, τα νομοθετικά όπως προέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Να αξιοποιήσει όλη την εμπειρία που αποκτήσαμε από την αξιολόγηση και την πρακτική εφαρμογή. Ε, νομίζω ότι όλοι επί της αρχής συμφωνούμε ότι θα καταθέσουμε την καλύτερη μας προσπάθεια. Ε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι το Κοινοβούλιο μας και με προηγούμενες εκθέσεις, επαναλαμβάνω, ε, με τον εξαίρετο συνάδελφο και πλέον ειδικό τον κύριο Κοέλιο, με όλα του τα κείμενα και τα ψηφίσματα, έχει ε, καθορίσει το επίπεδο στο οποίο κινείται και στο ίδιο υψηλό επίπεδο ευελπιστώ και εγώ να συνδράμω να κινηθούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Thank you. Having said Σας ευχαριστώ. Μετά από αυτά και με την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης που θα παρουσιαστεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΕ, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο σημείο 12 που αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Θα εξετάσουμε το σχέδιο ε, νομοδότησης και θα ληφθεί και απόφαση σε αυτή την κατάθεση τροπολογιών που θα επιβεβαιωθεί μετά από το πακέτο όσον αφορά την κατάσταση στην Νότιο Μεσόγειο που δημοσιεύτηκε τον Μάη 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να ζητήσει σύνταξη μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία. Η δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή ζητήθηκε να συντάξει μια έκθεση γνωμοδότηση και έχουμε μια συντάκτρια αυτή τη έκθεση γνωμοδότηση την κυρία Φλότρο. Θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της και θα έχουμε κάποιο περιθώριο να κάνουμε κάποια σχόλια. Η κυρία Φλότρο έχει τον λόγο λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσίαση αυτής της ε, μικρής ε, σε όγκο έκθεσης ε, διότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 1500 χαρακτήρες πάνω σε ένα τόσο δύσκολο και περίπλοκο ζήτημα να μπες τόσο περί τίνος πρόκειται μετά από τα λαϊκά κινήματα στο νότιο τμήμα της Μεσογείου η Κομισιόν συνέταξε μια σειρά ανακοινώσεων από το Μάρτιο λοιπόν υπήρξαν τρεις ανακοινώσεις δύο στα τέλη Μαΐου μία εξ αυτών αφορά άμεσα τα θέματα που εξετάζουμε εδώ ως Επιτροπή, δηλαδή τα ζητήματα μετανάστευσης, κινητικότητας και ασφάλειας, δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, προσπάθησα μέσα στο έγγραφό μου να συμπεριλάβω κάποιες συστάσεις ε, προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εξάλλου θα έχω μια συνάντηση με τον εισηγητή Μάριο Νταβίδη σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ε, Νοτιού Μεσογείου έτσι ώστε να συμπεριθούν αυτά στο τελικό έγγραφο το οποίο θα παρουσιάσει ο συνάδελφο ΣΥΔΙΕΚ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Λοιπόν, ε, επικεντρώθηκα σε ζητήματα κινητικότητα, ε, μετανάστευση το σύντομα καθώς ε, το, τα νέα δεδομένα αναφέρουν ότι τα επεκτενόμενα στην Νότιο Μεσόγειο μας ε, εγκαλούν για ε, μετά από την πολιτική που ασκήθηκε μέχρι την έναρξη των κινημάτων, εξεγέρσεων κλπ. και να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της πολιτικής ε, καταστολής που εφάρμοσαν ε, πολλά οι ηγέτες ε, του Νότου Μεσογείου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε παραπέρα και να σκεφτούμε τα ζητήματα της κινητικότητας και της μετανάστευσης ανάμεσα στις δύο όχθες Μεσογείου. Κάτι το οποίο αναφέρω στο κείμενό μου ως win-to-win win to win situation, δηλαδή όπου όλες οι πλευρές θα βγουν κερδισμένε. και θεωρούμε ότι το δικαίωμα στην κινητικότητα θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα δικαίωμα θεμελιώδες ε, του ανθρώπου που αποτελεί κομμάτι της ε, δημοκρατίας και του εκδημοκρατισμού μαζί με το δίκαιο στην αξιοπρέπεια και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 1 των προτάσεών μου. Θα ήθελα να ζητήσω να αναρωτηθούμε σχετικά με το σύνδεσμο ο οποίος γίνεται πολύ συχνά και στην ίδια μας την Επιτροπή όπου ε, ε, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα θετικές ε, τουλάχιστον στον τομέα της κινητικότητας αυτή η αλληλεξάρτηση λοιπόν, το οποίο διεκδικεί πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νόμιμη μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, υπογραφή συμφωνώ και λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε αυτή την αλληλεξάρτηση, να την αξιολογήσουμε όπως η Κομισιόν αξιολόγησε τις ε, συμφωνίες ε, επανεισδοχής ε, που είχαν διαπραγμάτευση και εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα δείτε λοιπόν και εσείς όπως και εγώ ότι αυτή αυτές οι εκθέσει δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά και η Κομισιόν παρά τα αυτά περιλαμβάνει το πακέτο τη νόμιμη μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης κλπ. Και, και θεωρεί ότι η νόμιμη μετανάστευση θα αποτελέσει ένα είδος ανταμοιβή για τις καλέ υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ελέγχου της παράνομης μετανάστευση. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα. Ε, εν πάση κρίνω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να περάσουμε σε αξιολόγηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρω στην παραθυπαρθών 3. Τώρα με κάποια μεταφραστικά προβλήματα και θα θέλω να αναφερθώ σε δύο και θα θέλω να διευθυνθούν τώρα. Το δίλημα της ε, αξιολόγησης να, αλλάξει και να ε, συμπεριληφθεί όρος κριτήρια. Τώρα ε, για τη χρηματοδότηση σχεδίων ε, για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών θα, είπα, δεν έλεγα ότι καλούμε την Κομισιόν να δώσει κατά προτεραιότητα κάποιες δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών προκειμένου να μην ε, εφαρμόσουν προγράμματα τα οποία δεν θα στήριζαν τα δικαιώματα των μεταναστών τουλάχιστον αναφέρομαι στο γαλλικό κείμενο αυτό λοιπόν θα μπορούσε να διαφωτίσει κάποιους, ε, κάποιους προβληματισμούς ε, τώρα. Η παράγραφος 6 είναι πολύ σημαντική, αφορά άλλους τομείς δράσης που δεν συνδέονται μόνο με τη που πρόκειται ένα μηχανισμό για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών ε, στην εφαρμογή αυτών των στόχων και των κριτηρίων και κατά την αξιολόγηση, διότι σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας είναι ένα θεμελιώδη στοιχείο, κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και την ε, αξιοπιστία μιας πολιτικής ε, που θέλει όλο και περισσότερα, να έχει δηλαδή τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση, άρα η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστική σημασίας. Εξάλλου ο κύριος Λεόν ε, ο οποίο ε, προλίγου μίλησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Επιθέσεων, φαίνεται ότι συνενεί με αυτή την προσέγγιση. Στην παράγραφο 3 ξέχασα να σα πω ότι θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως κάνει και ο Μάριο Νταβίντ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρξει μια απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων, μια ζώνη ελεύθερη προξενικών θεωρήσεων, μια πολιτική λοιπόν η οποία θα είναι πιστική και να την υλοποιήσουμε. Θεωρώ ότι με μια χώρα όπως η Τινησία μπορούμε να προχωρήσουμε με βάση αυτή την προοπτική. Και τέλος για να ολοκληρώσω επί του συνόλου των τραγικών γεγονότων που επηρέασαν ε, τα μεταναστευτικά κινήματα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Λιβύη και που προσέφυγαν είτε στην, στην Αίγυπτο είτε στην Ισία και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους ε, και δεν έχει υπάρξει η εγκατάστασή τους ε, τουλάχιστον ε, προς το παρόν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι έρευνες που γίνονται σχετικά με τα πλοιάρια των μεταναστών που να βάγισαν ε, και αυτό το αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν τη ζωή τους, να πνιγούν στη Μεσόγειο, αλλά και ε, διάφορα σκάφη τα οποία έφεραν ε, σημαία των ευρωπαϊκών κρατών μελών, τα οποία έπλεαν στην περιοχή, δυστυχώς δεν βοήθησαν τους, τα, τους ανθρώπους σε αυτά τα ναυάγια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες έρευνες, ανακρίσεις, διότι δεν εφαρμόστηκε η Συμφωνία Αναζήτησης και Διάσωσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στη συμφωνία που συνδεθεί ανάμεσα στις ε, Ιταλικές Αρχές και το Μεταβατικό Συμβούλιο, το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο τη Λιβύης. Είχα θέσει το ερώτημα στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι δεν έλαβε ποτέ γνώση ύπαρξη μια παρόμοια ε, συμφωνίας. Έθεσα το ερώτημα και σε άλλους συνομιλητέ. Ε, ίσως θα χρειαστεί εδώ να βρούμε μια διατύπωση που θα δείχνει ότι αυτή η συμφωνία δεν ε, έγινε γνωστή στο κοινό ούτε στα κοινοβούλια. Ως εκ τούτου εδώ υπάρχει έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας. Στηρίζομαι λοιπόν στις ε, τροπολογίες σας ε, για να βελτιώσω το κείμενο. Εγώ περιορίζομαι στα 1500 λέξεις ενώ οι τροπολογίες δεν έχουν αυτόν τον περιορισμό. Θα φροντίσω λοιπόν να τροποποιήσω καταλήλως το κείμενό μου. Και αυτή τη στιγμή την δίκον ους. Now, Πρόεδρος, να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αντίδρασή της και από την Προεδρία του Συμβουλίου. Πρωτού αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των μελών. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, κύριος Τζοβάνι Κρεμονίνη, παρακαλώ. Βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Fact, uh, Παρακαλώ. Uh, the... Ευχαριστώ. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωματικής Δράσης, Εξωτερικής Δράσης, όχι από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξεκινήσω λέγοντας ε, κάποια πράγματα και να δοθεί ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιο εξειδικευμένες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά θέματα μετανάστευσης κτλ. Θα ήθελα απλά να πω ότι τις παρατηρήσεις που έγιναν από την κυρία Φλότρο και νομίζω ότι έχουν τη σπουδαιότητά τους με ιδιαίτερο τρόπο. Ξεκινήσαμε ήδη με την εφαρμογή, την υλοποίηση των θεμάτων της ανακοίνωσης για μια νέα προσέγγιση για την αλλαγή στα θέματα γειτονίας, μια νέα σχέση γειτονίας, ιδιαίτερα όσον αφορά δημοσιονομικά κονδύλια τα οποία θα κινητοποιηθούν και θα διατεθούν θα υποβάλουμε επίσης μια νέα, ένα νέο σχέδιο κανονισμού μέχρι τα τέλη του έτους που θα δώσει τη δυνατότητα να ενισχυθεί ακόμα, να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο το θέμα των αρχών στην ανακοίνωση ενισχύοντας ε, τα θέματα πολιτικής ε, και χρηματοδότησης. Το θέμα της ε, νέας διαμόρφωσης αυτών των κοινωνιών είναι πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζετε προετοιμάζουμε μέσω για τη διευκόλυνση της κοινωνίας των πολιτών μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Αυτό το μέσο θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του 2012. Θα έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό 22 εκατομμυρίων ευρώ γενικά σε σχέση με αυτή την νέα προσέγγιση που θα πρέπει να εντάσει την κοινωνία, τη νέα κοινωνία σε βάθος όσον αφορά και την ίδια την εποπτεία αυτής της ε, νέας πολιτικής ε, γειτονίας από πλευράς Ευρώπης θα επεκτείνεται σε σχέση με τα θέματα αυτά της κοινωνίας. Θα ζητάμε από την κοινωνία να υπάρχει, να δώσει τοποθετήσεις και όσον αφορά τις ε, προτάσεις αυτές μέσω τακτών επαφών που θα υπάρχουν. Αλλά καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας διαφρομένος, δομημένος διάλογος με αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο για τη δημοκρατία μας που είναι ακριβώς για τους πολίτες αυτό, για τις οργανώσεις ε, που μπορούν να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των πολιτών και να προαγάγουν τη δημοκρατία για τα θέματα της μετανάστευσης ο συνάδελφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο εξειδικευμένα θα μπορέσει να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Φραντσέσκο Λουτσάνι το όνομά μου από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Home Affairs. Ε, πολύ σύντομα θα μπορούσα μόνο να σχολιάσω την παρουσίαση που έγινε από την κυρία Ευρωβουλευτή Φλότρο, εκφράζοντας πρώτα την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τις θετικές μελλοντικές αυτές επιτυχές ε, της ανακοίνωσης που έγινε τον Μάιο και που θα ισχύσει στο μέλλον και σε σχέση με την 24η Μαΐου για την έναρξη ενός διαλόγου όσον αφορά την κινητικότητα και τα θέματα μετανάστευσης στην νότια στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή η ανακοίνωση ως τμήμα αυτού του πακέτου, πακέτου πραγματικά είχε στόχο να, ανοίξει, να διανοίξει νέες δυνατότητες για την κινητικότητα και την μετανάστευση για τους πολίτες ε, της νότιας όχθης ε, της Μεσογείου που θα εμπλεκόντουσαν σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων και μέσα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρούσαν. Οι πτυχές ασφάλειας ε, που εντοπίστηκαν μας έκαναν να λάβουμε απαραίτητα στοιχεία υπόψη ως τμήμα αυτής ε, της συνεργασίας και διεργασίας. Όμως η κινητικότητα δεν είναι υποχρεωτικά ένα ε, αντι, αντιστάθμισμα που δίνεται όταν υλοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις αλλά είναι ο απότερος στόχος αυτής της συνεργασίας υπάρχει μια σταφής διασύνδεση μεταξύ ενός αριθμού θεμάτων που πρέπει να σημειώσουν πρόοδο υπό διαφορετικές πτυχές. Όμως, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτές τις δύο ανακοινώσεις, είναι μέσα σε ένα ανοιχτό πλαίσιο και είναι πολύ καινοτόμα αυτή η τοποθέτηση και νομίζω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω άλλες πτυχές. Μπορώ να ολοκληρώσω όμως λέγοντας ότι Επίσης ε, καλωσορίζουμε την πρόσκληση να υπάρξει ένας ε, διαρθρωμένος διάλογος με τις αρχές των τρίτων χωρών και αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα ανέλαβε πρωτοβουλία να έρθει σε επαφές ε, με τις αρχές εκείνων των χωρών που είχαν εντοπιστεί και είχαν προταθεί από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδιαίτερα την Ισία, Μαρόκο και Αίγυπτο. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή ήδη κατά τέλη Ιουνίου. Οι απαντήσεις, οι αντιδράσεις δεν ήταν άμεσα κάποιου χειροπιαστού χαρακτήρα. Δεν θα έλεγα δεν ήταν θετικές οι αντιδράσεις, οι πρώτες τοποθετήσεις. Οι αρχές όμως αυτών των χωρών ζήτησαν να υπάρξει ένας χρόνος περισυλλογής για να τα εξετάσουν αυτά τα θέματα. Ιδιαίτερα την Ισία και Αίγυπτος εμπλέκονται σε ένα πολύ σύνθετο ακαθόδες ε, ε, θέμα διεργασιών. Έχουμε σημαντικές εκλογές ε, που αναμένεται να διεξαχθούν και το Σεπτέμβριο, τον επόμενο μήνα και δεν ήταν εφικτό να καθοριστεί σχετική ημερομηνία για αυτόν τον διάλογο, την ένταξη του διαλόγου. Όμως είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον διάλογο. Φυσικά στο τεχνικό επίπεδο πολλές επαφές έχουν ήδη ε, προετοιμαστεί και προετοιμαζόμαστε για αυτό το έργο να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα κάποια, κάποιους ευρωβουλευτές που επιθυμούν να παρέμβουν. Θα έλεγα πρώτα να ακούσουμε όμως την από πλευρά Σίβιεκ που είναι εισηγητή για την Επιτροπή, ο κύριο Μάρεκ Σίβιεκ, ο ε, εισηγητή τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, ο κύριο Σίβιεκ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για το έργο που επιτελέστηκε από την κυρία εισηγήτρια, την κυρία συντάκτρια γνωμοδότηση, την κυρία Φλότρα. Κυρίως με αυτή τη, σε σχέση με αυτή την έκθεση θα ήθελα να σας πω ότι εμείς στην πολιτική γειτονία κάνουμε λόγο εδώ και έξι μήνες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα με την έκθεση από πλευρά του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα και τώρα εργαζόμαστε εμείς επί ενός θέματος που είναι μια απόδειξη χειροπιαστή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συγκροτήσει μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά την πολιτική γειτονία και έναντι της νότιας όχθης της Μεσογείου. Να έχουμε μια θέση. Στι 29 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί μια σύνοδος κορυφής στη Βασοβία για τις σχέσεις με την Ανατολική Συνιστόσα. Έχουμε όμως ένα ευρύτερο πλαίσιο τη πολιτική γειτονία ούτως ή άλλω. Θέλω να αφαιρθώ σε αυτά τα θέματα και σε σχέση και με την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών που, ε, και να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Αλλά αν επιτρέπετε θα ήθελα να πω ότι η συντάκτρια γνωμοδότησης και εσείς θα πρέπει να δείτε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης και της έκθεσης. Κάνουμε λόγο για ένα συνολικό πλαίσιο μιας πολιτικής γειτονίας. Κάνουμε λόγο για τις νέες πραγματικότητες, πολιτικές και κοινωνικές στο βορρά της Αφρικής, στη βόρεια όχθη της Αφρικής, νότια όχθη της Μεσογείου τι θα κάνουμε με την πολιτική γειτονία στο ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πολιτική παρότι αφορά διαφορετικά γεωγραφικά τμήματα να έχει κοινά χαρακτηριστικά και πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, πού θα τονίσουμε, πού θα ενδυναμώσουμε ε, κάποια από αυτά και πού θα θέσουμε το κέντρο βάρους. Ο δημοκρατισμός είναι σημαντικό θέμα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολλαπλές επαφές με την κοινωνία των πολιτών, η υποστήριξη της κοινωνίας σφαιρικά και, στην, ε, και των οργανώσεων των πολιτών. Αυτά είναι, όπω προανέφερα, χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν και να χαρακτηρίζουν τι σχέσει που θα διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σχέσει τη με αυτές τις χώρες. Θεμέλια ισχυρά και να μην εξαρτάται από την βούληση ενό ή άλλου. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτέ τι χώρε και που επιθυμούν να θεμελιώσουν νέε σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τι θεμελιώσουν σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε μέσα σε αυτά τα θέματα να προαγάγουμε. Αυτό υπενθυμίζουμε σε σχέση με αυτά τα θέματα. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο σχέδιο για το οποίο κάνετε εσείς λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα οποία αναφέρονται στο σημείο 6 και αυτά τα οποία αφορούν την ύπαρξη και υποστήριξη αυτής της νέας πολιτικής. Κάνω λόγο για έναν μηχανισμό εποπτείας, επίβλεψης η επόπτευση και για τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών με τα benchmarks, τι βέλτιστες προδιαγραφές, με τακτικές επαφές με τις ελίτ, με τους νέους. Είναι πολύ καλά όλα αυτά και αν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα θα σημειώσουν πρόοδο και θα σημειώσουν σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό που όπως πιστεύω εγώ είναι κάτι στο οποίο επικεντρώνεστε εσεί ω ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τα θέματα κινητικότητα και μετανάστευση αυτά και επίσης του σεβασμού των δικαιωμάτων από την άλλη όμως πλευρά και το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λοιπά. Εφιστώ την προσοχή στο εξή για την πρόταση που υλοποίησε και υπέβαλε ο Μάριο Νταβίδ. Αυτό το θέμα είναι αδιαμφισβήτητα ως, έχει ως εξή. το άρθρο 21 από πλευράς ε, ε, εισήγηση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να σταματήσει, να πάψει να ισχύει ε, το καθεστώς θεωρήσεων διαβατηρίων. Αυτό είναι ο στόχος μας, απότερος στόχος μας, διότι οι θεωρήσεις διαβατηρίων σε σχέση με τις σχέσεις που θέλουμε να έχουμε με αυτές τις χώρες, θέλουμε σίγουρα να είναι σεβαστά τα δικαιώματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι οι θεωρήσεις διαβατηρίων πρέπει να ανήκουν πια στο παρελθόν, πρέπει να τις ξεπεράσουμε πια και ε, κινητικότητα όσον αφορά την ορολογία όπως χρησιμοποιείται δεν είναι μόνο να διευκολυνθεί η εισαγωγή εργατικών χεριών. Όχι. Αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο εδώ είναι η ροή, οι μεταναστευτικές ροές μεταξύ κοινωνιών. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από το εργατικό δυναμικό, από τα χέρια, από το ε, ε, δυναμικό των εργαζομένων. Όλοι εκείνοι που θέλουν ε, να προσέλθουν λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενοι μια ολόκληρη σειρά αρχών, τότε είναι ευπρόσδεκτη. Για εκείνους που θέλουν και μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν εδώ και έχουν και την έγκριση της χώρας που τους προσκαλεί, είναι μια ανοιχτή διαδικασία για τους νέους. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια, κυρία Φλότρ, και αναμένουμε την τελική έκδοση αυτής της έκθεσης. Το πρόγραμμα είναι μέχρι τα τέλη του έτους να μπορέσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο να ολοκληρώσουμε και να έχουμε τις τελευταίες συστάσεις για την πολιτική γειτονία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά και την Ανατολική Συνιστόσα και τον Νότο. Ευχαριστώ. Ανοίγουμε τώρα τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Νεντέλτσεβα, έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Φλότρου για την γνωμοδότησή τη, η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να ευχαριστώ επίση για την παρουσίαση που μα έκανε. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία έχει ανάγκη από ανανέωση και θα χαίρομαι που μπορούμε να εξετάσουμε σήμερα το ζήτημα μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις ιδιαίτερα στους γείτονές μας του Αγίου. Θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των δημοκρατικών αρχών και την έννοια του δικαιώματος στην κινητικότητα. Τώρα για τις δημοκρατικές ε, ε, αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι στην Επιτροπή μας ΛΥΜΠΕ είμαστε καρεξοχήν Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα αυτό. Είναι δική μας αρμοδιότητα και ο ε, τίτλος του παραγράφου 1 θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι απαιτητική για να μην πούμε αδιάλακτη απέναντι στους εταίρους της σε ζητήματα δημοκρατικών αρχών. Χρειάζεται επίσης να αναφέρουμε τη σημασία των ελεύθερων εκλογών, την, ε, σεβασμό ε, του δικαιώματο σε, σε συνάθρηση, σε κλπ. Θα πρέπει να έχουμε μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη που θα καταπολεμεί την διαφθορά και ε, δημοκρατικές αστυνομικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικές αρχές, προφανείς μεν, αλλά είναι αυτές οι αρχές που συχνά τις ξεχνάμε πιο περισσότερες φορές. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περαιτέρω. Αυτό είναι το πρώτο σημείο μου τώρα για το δεύτερο το θέμα το δικαιώματο στην κινητικότητα. Θα ήθελα να εξετάσουμε το ζήτημα με τον δυνατότερο ευρύ και πλήρη τρόπο. Να επενθυμίσουμε ότι αυτή η αρχή στην κινητικότητα υφίσταται, κάτι το οποίο πράτεται στην γνωμοδότηση, αλλά να επενθυμίσουμε ότι δεν είναι μονόδρομος και αυτό για δύο λόγους. θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι όταν οι εταιρικές σχέσεις γειτονία συνάπτονται θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Χρησιμοποιείται την πολύ σωστή διατύπωση προσέγγιση ε, win-win. Θα ήθελα να τονίσουμε ότι η κοινωνικότητα αποτελεί μια ανάγκη οικονομική για δύο πτυχές, πλευρές, αλλά ε, ενέχει το κίνδυνο της ε, διαφυγής εγκεφάλων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα χρειάζεται να οδηγήσουμε μια χώρα στην εγκατάλειψη εγκεφάλων, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα βοηθάει την ε, επιστροφή των ε, προσώπων αυτών, ιδιαίτερα των ερευνητών και των φοιτητών. Αυτή η κοινωνικότητα, λοιπόν θα με σημαίνει ε, λευκή επιταγή προς όλους και να επιτρέψουμε την, και να, να υπάρξει καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ε, κλπ. Αυτά θα πρέπει να είναι πτυχές που αναφέρονται στην έκθεση, όπως επίσης και το ζήτημα της ενίσχυσης ε, της δυνατότητας διαχείρισης των συνόρων ε, και τη συνεργασία ανάμεσα στις νομικές αρχές. Αυτά ήταν δύο σημεία που ήθελα να θίξω και ευχαριστώ για μια ακόμα φορά την κυρία Φλότρο για την εξαιρετική εργασία της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Μίλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο ερώτημα προς τον συγκητή αλλά προς την Κομισιόν. Ήμουν πρόσφατα σε μια χώρα που γειτονεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει συμφωνία βίζας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ρώτησαν γιατί ο Ισημερινός και η Κωνσταντίνα και οι πολίτες τους δηλαδή μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο για μια χώρα που γειτονεύει. Μπορεί η Κομισιόν να μου εξηγήσει υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι χώρες για να έχουν ε, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα ή γίνεται σε βάση ad hoc. Τι συμβαίνει, τι να πω σε μια χώρα που με ρώτησε γιατί δεν μπορούν οι πολίτες μου να πάνε ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Κύριος ε, Τριανταφλίδης Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τον συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Φλότρ για το εξαιρετικό της έργο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ανακοίνωσής της, νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει, προσπαθεί να αντιδράσει γρήγορα σε σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο άμεσο περιβάλλον ε, περιβάλλον της ε, σε χώρες με τις οποίες είμαστε σε στενή συνεργασία εδώ και δεκαετίες και προσπαθεί να βρει μια συνεκτική πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει όλες τι πτυχέ, όπως παραδείγματο χάρη η τη της δημοκρατίας, εμπόριο, οικονομική ανάπτυξη, μετανάστευση και έλεγχος των συνόρων κτλ. Όμως μου φαίνεται πως αυτό το οποίο προτείνεται δεν είναι μια νέα απάντηση αλλά μια διαρθρωμένη λίστα των όσων κάνει ήδη εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε πως αυτά δεν λειτουργήσαν. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι γνήσιες εταιρικέ σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις για να προωθηθεί ευημερία όλων των μερών της κοινωνίας. Οι όροι δεν θα πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της Ένωσης, τις χώρες αυτές, αλλά με τους στόχους που οι, χω... κάτοικοι της εν λόγω χώρας θέλουν να επιτύχουν. Αυτό σημαίνει το να νιώθουν δική τους την πολιτική. Αυτό σημαίνει βαθιά δημοκρατία και αυτό σημαίνει και πολυμορφία. Η πολυμορφία δεν αφορά μόνο την συνύπαρξη διαφορετικών λαών και πολιτισμών σε ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά και να αποδεχτούμε πως διαφορετικά μοντέλα πολιτικής διακυβέρνησης και οικονομική οργάνωση, είναι βιώσιμα ακόμα και υποφελή αρκεί να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του α, λόγω πληθυσμού. Εάν είναι να χρησιμοποιούμε λέξεις και τέτοια συνθήματα όπως βαθιά δημοκρατία και ποικιλομορφία πρέπει να έχουν κάποια ουσία, αλλιώς δεν σημαίνουν τίποτα. Και νομίζω πως αυτό ακριβώς κάνει η ΕΛΕΝ στη γνωμοδότησή της μέσω συγκεκριμένων προτάσεων. Στηρίζουμε την πρότασή της και σκοπεύουμε να υποβάλουμε κάποιες συμπληρωματικές τροπολογίες για να αναφερθεί η ανάγκη να ερευνηθεί η συστηματική επαναπροώθηση στην ε, την Ισία καθώς επίσης και η παράληψη, η διάδοση, στην, διάσωση στην θάλασσα από κάποια κράτη και πλοία του ΝΑΤΟ και να υπενθυμίσουμε και να ζητήσουμε από την ε, Ιταλική κυβέρνηση το κείμενο της συμφωνίας με την, την Ισία. Σας ευχαριστώ κύριος Μπρόγκς. Ναι, ακούσαμε απόψε πως οι εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική θα ε, οδηγήσουν και πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κινητικότητα και μετανάστευση. Το αντίθετο πρέπει να συμβεί, φαντάζομαι, καθώς γίνονται λιγότερο καταπιεστικά αυτών των καθεστών, τα καθεστώτα αυτών των χωρών, θα πρέπει να μην υπάρχει ανάγκη να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη οι μόνοι οι οποίοι θα βρουν δυσάρεστη την ατμόσφαιρα στη Λιβύη είναι η οικογένεια και οι φίλοι του κυρίου Καντάφ. Φαντάζομαι θα είναι πρώτος που θα ζητήσει άσυλο. Πολλές χιλιάδες ζωών χάθηκαν στις ε, συγκρούσεις στη Λιβύη και κάποιοι θεωρούσαν πως ο στόχος ήταν να γίνει η Λιβύη καλύτερο μέρος για να ζει κανείς και όχι για να φύγει. Ίσως όλα αυτά είναι παραδοχή του ότι όποτε η Δύση ανακατεύεται σε χώρες ε, στις οποίες δεν έχει καμία δουλειά, αφήνουν τις χώρες αυτές, όπως το Ιράκ, με περισσότερα προβλήματα και περισσότερη καταπίεση και όχι λιγότερα. Σας ευχαριστώ. Τώρα, έγιναν κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ε, συγκεκριμένα, οπότε προτείνω η εκπρόσωπος της Κομισιόν, εάν έχει να δώσει κάποια απάντηση, να το κάνει τώρα. Ποιος θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν, παρακαλώ. Ε, τέθη ένα ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια βάσει τα οποία οι διάφορες χώρες ε, ε, εφαρμόζουν για την ε, ε, χορήγηση θεωρήσεων. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο. Παρακαλώ κύριε Ντεκώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι παρόν για το επόμενο σημείο που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού 539-2001. Και αυτό αφορά τον αρνητικό κατάλογο και τον θετικό κατάλογο, δηλαδή τις χώρες ε, των οποίων οι απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Λοιπόν, απαντώντας ε, στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθη αναφορικά με κριτήρια, θα περιοριστώ σε αυτό το στάδιο να παραθέσω τα κριτήρια όπως ε, τα έθεσε ο ενωσιακός νομοθέτης στο προνόμιο αυτού του κανονισμού 539-2001 και παραθέτω αποτελεσματικότητα αυτών των κρατών των οποίων οι πίκο υπόκεινται στην έκδοση ε, θεώρησης και ε, χωρών που, των πικών που απαλλάσσονται εξετάζονται κατά περίπτωση με βάση μια σειρά κριτηρίων που ε, άπτονται ε, μεταξύ άλλων στην παράνομη μετανάστευση, την ε, δημόσια πολιτική ασφάλειας ε, και στις σχέσεις ε, με τις τρίτε χώρες και επίσης ε, δίνεται σημασία στο θέμα της αμοιβαιότητας και της περιφερειακής συνοχής. Έχουμε λοιπόν πέντε βασικά κριτήρια. Φυσικά δεν πρόκειται για μαθηματικά, μιλάμε για πολιτικές αξιολογήσεις και πολιτικά κριτήρια τα οποία γίνονται και δεν είμαι σίγουρος ε, σε ποια γειτονική χώρα αναφέρονταν ο αξιότιμος κύριος ε, βουλευτής αλλά ε, η λίστα που σας ανέφερα έχει όπως σας είπα τουλάχιστον έτσι είναι διατυπωμένη σήμερα και πέρυσι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να περάσουν Κάποιε χώρε από την αρνητικό κατάλογο στην θετικό κατάλογο με βάση τα κριτήρια που προανέφερα. Και τέλος, αυτοί οι κατάλογοι τακτικά αναθεωρούνται διότι τα κριτήρια και οι συνθήκες αλλάζουν και νέες αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνουν σε τακτά διαστήματα. Ευχαριστώ. Ωραία. Και τώρα η κυρία Φλότρο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο και σχολίασαν, ε, θα περιμένω τις τροπολογίες τους. Ε, πιστεύω ότι η απάντηση που μόλις μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Τροπή καταδεικνύει ότι η σημερινή προσέγγιση της πολιτικής ε, γειτονία και μετανάστευσης δεν ε, στηρίζεται στο γεγονό ότι οι χώρε αυτές είναι γειτονικέ. Αυτά τα οποία ισχυρίζεστε ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου. Εμείς εδώ θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα είναι αφιερωμένη στις γειτονικέ χώρες οι οποίες γνωρίζουν την δημοκρατική μεταλλαγή και φορά φυσικά τους ε, μετανάστες που ζουν στις χώρες μας και τα παιδιά μεταναστών. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, να είμαστε πιο ανοιχτοί και φυσικά αυτό με βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν στα τέλη Μαΐου. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε παραπάνω για να χαράξουμε ένα νέο δρόμο για μια ζώνη ελεύθερη θεωρήσεων όπου θα υπάρχει μια υπεύθυνη μετανάστευση διότι αυτή η μετανάστευση είναι μάλλον με τρόπο άναρχο, φωνικό θα έλεγα και θέτει τους ανθρώπους σε επισφαλή κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να χαράξουμε ένα δρόμο για μια κινητικότητα win-win όπως επανειλημμένα αναφέρθηκε. Περιμένω λοιπόν ε, τις προτάσεις σας επί των σημείων Ο κύριος Σίβιατ ε, μας κάλεσε να εξετάσουμε τον σφαιρικό χαρακτήρα της έκθεσης. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επειδή έχουμε κάποια συγκεκριμένα όρια που μας έχουν τεθεί στο πλαίσιο λοιπόν της ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι σε ζητήματα κινητικότητας και μετανάστευσης και τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του. Δεν συμφωνώ με την άποψή του αναφορικά με την κινητικότητα που δεν θα πρέπει να ανταποκρίνεται με μια ικανότητα μετανάστευσης ε, νόμιμης, ε, νόμιμου εργατικού δυναμικού. Θεωρώ ότι όλοι κρίνουν πως η Ευρώπη θα έχει όλο και, ανάγκη όλο και περισσότερους ε, μετανάστες, εργατικά χέρια λοιπόν και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα, θα προσφέρει πλούτο τόσο σε εμάς ως Ευρώπη όσο και στις χώρες καταγωγής. Για μένα λοιπόν το δικαίωμα στην κινητικότητα είναι και η δυνατότητα όντως ε, της ε, μετανάστευσης ε, μιας μορφής εργασίας εξελιγμένης και όχι επισφαλούς. Θα τα ξαναπούμε όποτε το επιθυμείτε και αυτό με βάση τις προτάσεις που θα μου Ευχαριστώ. ευχαριστούμε κυρία Φλότο. Τώρα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτό που έχει τεθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έτσι, η δική μας Επιτροπή θα πρέπει στις 17 ε, Οκτωβρίου να ψηφίσει. Ακριβώς λόγω αυτού προτείνουμε η προθεσμία και κατάθεση τροπολογιών να καθοριστεί 14 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. 14 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Στις αρχές Οκτωβρίου πρωτού ψηφίσουμε θα συζητηθούν αυτές οι τροπολογίες στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Περνάμε στο σημείο 13. 13. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου καθορίζοντας ε, τις τρίτες χώρες ε, οι υπήκοοι των οποίων πρέπει να έχουν θεώρηση διαβατηρίων διασχίζοντας τα εξωτερικά σύνορα και τον κατάλογο εκείνων που απαλλάσσονται από αυτές τις υποχρεώσεις. Έχουμε ως στόχο τη συζήτηση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας εισηγητή τον συνάδελφο Δίας Μέρα. Να υπενθυμίσω απλά και μόνο ότι Αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά ρυθμίσεις που έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Πρόσφατες τροποποιήσεις που επικεντρώθηκαν στην αναθεώρηση και του θετικού και του αρνητικού καταλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων όσον αφορά τον κανονισμό και υπάρχει ανάγκη περαιτέρω τεχνικών τροποποιήσεων καθώς επίσης και επί του κυρίου κειμένου ενισχύοντας την νομική βεβαιότητα με κανόνες για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν καλυπτόντουσαν από τον κανονισμό, προσαρμόζοντας κάποιους ορισμούς προς αυτό το στόχο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Τζάντε Κόιστερ είναι από ό,τι γνωρίζω ο εκπρόσωπος και μετά από τη δική του παρουσίαση θα αρχίσει η συζήτηση με την παρέμβαση του εισηγητή πρώτα κύριου Μέρα. Κύριε λοιπόν εκπρόσωπε της Επιτροπής έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το στοιχείο πυρήνα αυτού του κανονισμού 539 του 2001 φυσικά είναι όπως αποκαλείται ο θετικός και ο αρνητικός κατάλογος που μόλις προαναφέρθηκαν. Αυτά είναι τα, η ακρογωνιαίοι λύθη της ε, σημερινής πολιτικής θεωρήσεων διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως αναφέρθηκε αυτοί οι κανονισμοί, αυτοί οι κατάλογοι έχουν σε τακτά διαστήματα προσαρμοστεί και ε, επικαιροποιηθεί και είχε το λέγει του το κοινοβούλιο κατά τα τελευταία ε, χρόνια Επίσης ε, η τροποποίηση των διατάξεων αυτού του κανονισμού ε, είχε εξεταστεί. Με μια πρώτη ματιά αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα τεχνικό καθαρά θέμα και στην πρόταση που θα παρουσιάσω τώρα υπάρχουν πράγματι κάποιες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες για τις οποίες το κείμενο του τρέχοντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα θέματα μεγάλης πολιτικής σπουδαιότητας και όχι κατελάχιστον και η ρήτρα διασφάλισης ή δικλίδα ασφαλείας που θέλει να εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό 539 που θα επέτρεπε μια απλουστευμένη διαδικασία ώστε να καταργηθεί η απαλλαγή ε, θεωρήσεων διαβατηρίων για μια τρίτη, συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρόνο έχω πρόεδρε για να παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Αν δω το πρόγραμμα της ημερήσιας διαταξής σας υπάρχει όμως μια πρόταση που θα ήθελα ούτως ή άλλως να κάνω μια παρατήρηση και αυτή είναι να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που ακολουθούσαμε και σε σχέση με άλλες προτάσεις όσον αφορά τα, τους ελέγχους συνόρων και ε, σε σχέση και με ε, τις θεωρήσεις διαβατηρίων, σε σχέση με μια τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση με τον εισηγητή Σιώδη, εισηγητές και άλλους που θα ενδιαφερόντουσαν, όπου λεπτός θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε πάσης φύσεως ερωτήματα και στα πιο τεχνικού χαρακτήρα χωρίς να στρεβλώσουμε τη συζήτηση στην επίσημη συνεδρίασή σας τώρα. Θα μπορούσα να προσφέρω από πλευρά των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προθυμία μας να διεξαχθεί μια τέτοια συνάντηση μαζί σας. Εσείς θα αποφασίσατε αν είναι σκόπιμο και εποφελές να διεξαχθεί μια τέτοια συνάντηση μαζί μας. Εμείς είμαστε όμως πρόθυμοι. Περιορίζομαι λοιπόν, μια και ο χρόνος πιέζει, στο να επικεντρώσω την ε, ε, παρέμβασή μου στην δικλίδα, στη ρήτρα διασφάλισης ε, και για τους μηχανισμούς που προτείνονται κάποιες αλλαγές, κάποιες προσαρμογές που είναι τα πιο πολιτικά, από πολιτικής πλευράς σημαντικά τμήματα αυτής της πρότασης. Με τη ρήτρα διασφάλισης λοιπόν ξεκινώ ένα μηχανισμό ώστε προσωρινά να αρθεί η απαλλαγή διαβα... χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων όσον αφορά δηλαδή τον θετικό κατάλογο για κάποιες χώρες. Ίσως θα θεωρηθεί έκπληξη ότι υποβάλλει η πρόταση μια τέτοιου είδους ε, ρήτρα διασφάλισης, δικλίδα ασφαλείας για αυτό το μηχανισμό. Όμως η ίδια, η εμπειρία πέρυσι μας δίδαξε, τα βιώματα πέρυσι μας έδειξαν ότι <clears throat> μπορεί να δημιουργηθούν δυσκολίες σε κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να, είναι, να τύχει ε, κατάχρησης ε, μια τέτοια περίπτωση για ε, υπήκος μιας τρίτης χώρας. Η ιδέα της ρήτρας διασφάλισης δεν είναι καθόλου καινούρια σε όλες τις, ε, σε όλες τις ε, συμβάσεις και συμφωνίες και στην ε, συνθήκη Λισαβόνας έχουμε μια ρήτρα διασφάλισης ή δικλίδα ασφαλείας με απλουστευμένη διαδικασία για την υιοθέτηση μέτρων όπως εδώ την απαλλαγή όσον αφορά χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων για υπο... υπηκός χωρών. Υπήρχε λοιπόν και η πρόβλεψη αυτή της ένταξης ε, αυτής της ε, δικλίδας διασφαλείας. Έχει ε, καταστήσει στενότερο το φάσμα τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τα θέματα ασύλου. Και αυτή η δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας καθόλου δεν θίγεται από την ε, δικλίδα ασφαλείας που προτείνουμε εμείς σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα θεωρήσεων διαβατηρίων. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι συμπληρωματικός μηχανισμός στην δικλίδα ασφαλείας που προβλέπεται από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, περιοριζόμενη στον τομέα του, της χορήγησης ασύλου και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι σε αυτό το σημείο οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρας έκτακτης κατάστασης ε, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα απαλλαγής ε, δεν θα υπάρχει αυτοματισμός με κανένα τρόπο οποιαδήποτε διαδικασία υιοθετηθεί στο τέλος ε, για την πρόταση που θα υιοθετηθεί από τον συνομοθέτη. Πάντα μια αξιολόγηση θα πρέπει να προηγείται και όχι με αυτοματισμό. Αν μέτρα σε σχέση με την δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά συνθήκη θα υπαρκούν για να αντιδράσουμε και να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες όσον αφορά και τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων. Τα δύο αυτά λοιπόν θα είναι συμπληρωματικού χαρακτήρα μέτρα. Ένα πράγμα θα ήθελα να τονίσω Όσον αφορά την έγκριση αυτή τη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τύπο, αναφέρθηκαν κάποιε αναφορέ σε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, όπου οι πίκοοι αυτών των χωρών δημιούργησαν κάποια προβλήματα πέρσι. Θα είμαι κάθετο επ' αυτού. Αυτή δεν είναι μια πολιτική συγκεκριμένη για κάποιε χώρε ή για κάποιε περιφέρειες ή περιοχέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνουμε γενικού χαρακτήρα δικλίδα ασφαλεία, ρήτρα ασφαλεία. που χρονικά θα επέτρεπε να καταργηθούν οι απαλλαγές θεωρήσεων διαβατηρίων για τρίτες χώρες αν τα κριτήρια για, την, ε, ε, αυτή την ε, απέτηση θα υλοποιούνται. Και αυτό με οδηγεί στις διεργασίες, στη διαδικασία για αυτό το μηχανισμό ασφαλείας. Για να καταργηθούν οι απαλλαγές θεωρήσεων διαβατηρίων δύο διαδικασίες θα ήταν διαθέσιμες. Η πρώτη θα ήταν να ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία συναπόφασης όμως πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πλέον ότι κάτι τέτοιο δεν προσφέρει αναγκαστικά την δυνατότητα να έχουμε την ταχύτερη υιοθέτηση του μέτρου κατάργησης ε, αυτής της απαλλαγής. Θα έλεγα η συναπόφαση εξορισμού απαιτεί κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η άλλη όμως εναλλακτική λύση είναι να δώσουμε εκτελεστικές εξουσίες κατά εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρίσμα της αποκαλούμενης επιτροπολογίας. Και φυσικά στη συνέχεια τότε θα πρέπει να υπάρχουν απόλυτα εξειδικευμένοι κανόνες, συγκεκριμένοι κανόνες για αυτή τη διεργασία και σαφή κριτήρια που θα επιτρέπουν τη δρομολόγηση και λειτουργία αυτή τη ρήτρα διασφάλιση. Δεν θα σα παρουσιάσω όλε τι λεπτομέρειε αυτών των κριτηρίων σήμερα και τώρα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια έκτακτη περίπτωση όπου μια πιθανή κατάργηση των απαλλαγών θεωρήσεων διαβατηρίων θα έπρεπε να εξεταστεί. Όμως προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ποσοστοποιημένα κριτήρια που μπορούν να ε, δώσουν τη δυνατότητα να κρίνουμε τα σχετικά θέματα ακόμα και σε σχέση με τον αριθμό των παράνομα ε, υφιστάμενων πολιτών μιας τρίτης χώρας ε, που θα δικαιολογούσαν την δρομολόγηση αυτών των διεργασιών. Όμως όλα αυτά θα λειτουργήσουν από πλευρά των κρατών μελών. Αν και τότε όταν θα υλοποιούνται αυτά τα κριτήρια, όχι αυτόματα με αυτοποιημένο τρόπο, δεν θα καταργηθούν, ε, δεν θα υπάρξει απαλλαγή των θεωρήσεων διαβατηρίων αυτόματα, αλλά θα πρέπει πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι να κάνει μια αξιολόγηση, να εκτιμήσει αν η έκτακτη κατεπίγουσα κατάσταση που θα αντιμετώπιζε ένα κράτος και οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα έπρεπε να οδηγήσουν στο να ληφθούν και υπόψη τα στοιχεία της Frontex, της ΕΑΣΟ και των κρατών μελών κατ' όλα αυτά. Δεν θα υπάρχει λοιπόν αυτοματισμός και έτσι σε σχέση με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτών των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολύ προσεκτική μελέτη συγκεκριμένων στοιχείων. Θα πρέπει να αναγνωριστεί φυσικά ότι η επιτροπολογία δεν προσφέρει μεγάλο περιθώριο για παρέμβαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και από αυτού του σημείου θα θεωρούσα και θα έλεγα ότι πρέπει φυσικά να επιστήσω την προσοχή σας επί ενός σημείου επί του οποίου ε, τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επεξηγηματικό μνημόνιο. Μια σαφή πολιτική δέσμευση. Και αναφέρομαι ως παράθεμα. Θα ανταλλάξει απόψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν υπάρχει η πρόταση κατάργησης ε, της απαλλαγής θεωρήσεων διαβατηρίων για μία ή περισσότερες χώρες Είμαστε πρόθυμοι και έχουμε την βούληση να εξετάσουμε μαζί σα, με εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και πότε μια τέτοια πολιτική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επισημοποιηθεί και να δρομολογηθεί. Το Κοινοβούλιο υπό αυτό το πλαίσιο θα είχε μόνο το δικαίωμα εξέτασης, δηλαδή να εξετάσει και να δει αν με τα προβλεπόμενα ε, στοχευόμενα μέτρα η Επιτροπή ξεπερνά τις εκτελεστικές εξουσίες που της έχουν ανατεθεί ή όχι όλο και όλο αυτό. Δεν είναι όμως πλήρης εξουσίες να προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο αλλαγές και τροποποιήσεις επί των προβλεπόμενων αυτών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάργηση απαλλαγής θεωρήσεων διαβατηρίων για τους υπηκόους μιας τρίτης χώρας. Αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα επί του οποίου θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις απόψεις σας για τρόπους για να επισημοποιηθεί αυτή η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο Εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όπως προανέφερα ήδη, δεν υπάρχει αυτοματισμός σε αυτή τη διεργασία. Σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης ε, μετά από ειδοποίηση κράτους μέλους θα υπάρξει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή σχετικά στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη και την χρήση της δυνατότητας της ρήτρας διασφάλισης ε, δικλίδας ασφαλείας. Έχουμε πάλι εδώ την ίδια δηλαδή ρήτρα που προβλέπει ως ίστατη ε, ας το πω έτσι δυνατότητα αυτό το να καταργηθούν οι απαλλαγέ θεωρήσεων διαβατηρίων ως κατακλίδα. Και όσον αφορά τον μηχανισμό αμοιβαιότητας, πρόεδρε, δύο λόγια. Έχουμε ήδη ένα τέτοιο μηχανισμό με την απλουστευμένη διεργασία στον τρέχοντα υφιστάμενο κανονισμό. Αλλά αυτή η διεργασία δεν είναι συμβατή με τη συναπόφαση που εφαρμόζεται όσον αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων το 2004-2005 αποφασίστηκε αυτός ο μηχανισμός πριν από την εισαγωγή του μηχανισμού συναπόφαση. Εμείς προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η, διαδικασία ώστε να λαμβάνεται πλήρω υπόψη και να είναι σεβαστή η διαδικασία πλήρου συναπόφαση που εφαρμόζεται για αυτόν τον τομέα για πιθανά μέτρα κυρώσεων εις βάρος τρίτων κρατών όσον αφορά την ε, χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων για κάποιες χώρες που επιβάλλει όμως θεωρήσεις διαβατηρίων για άλλες χώρες, για μία ή περισσότερες άλλες χώρες. Υπάρχουν προτάσεις να υπάρξουν και άλλες αλλαγές ώστε αυτός ο μηχανισμός να καταστεί πιο αποτελεσματικός, πιο λειτουργικός. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός όσο έχει τώρα. Όμως φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη και είναι ευήκον ους να ακούσει και το Συμβούλιο και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν υπάρξουν κάποιες άλλες αλλαγές που θα μπορούσαν να, γίνουν ώστε το πλαίσιο αυτό να καταστεί πιο αποτελεσματικό. Και τέλος, Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλες, δεν θα έλεγα καθαρά τεχνικού χαρακτήρα θέματα, αλλά όσον αφορά το πλαίσιο για ε, ε, τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων Τούρκων υπηκών μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και υπό το πλαίσιο της νομολογίας του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπάρχει και η δυνατότητα της, α, ε, ε, του 539 όσον αφορά τον κώδικα θεωρήσεων διαβατηρίων. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα θέματα που αξίζει να εξεταστούν περισσότερο σε βάθος μέσα στο πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης. Σαν συμπέρασμα επαναλαμβάνω την προσφορά μου προς εμάς. Να έχουμε μια τέτοια έκτακτη συνάντηση όπου θα συζητήσουμε πλήρως σε βάθος όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον εισηγητή. Ακούσαμε την παρουσίαση, λοιπόν θα ακούσουμε τώρα και την Πολωνική Προεδρία πριν μιλήσει ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της Επιτροπής. Ε, να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία ακούσαμε από την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα λέγομαι Φιλίπ Λισινσκή και είμαι αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Θεωρήσεων στο Συμβούλιο. Να σας πω λοιπόν πως είχαμε ε, την πρώτη άμεση ανταλλαγή απόψεων και την πρώτη ανάγνωση της πρότασης της Κομισιόν στην Ομάδα Εργασίας μας και μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει μεγάλη απόκληση απόψεων μεταξύ των αντιπροσώπιών. Σε μεγάλο βαθμό τα βασικά σημεία της πρώτης κομισιόν αντιμετωπίστηκαν με κατανόηση και ελπίζω να μην προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία θα θέλαμε να επανέλθουμε. Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το πώς τα κριτήρια μιας πιθανής εισαγωγής ε, του μηχανισμού διασφάλισης ή άρσης ε, θα λειτουργήσουν και βεβαίως θα πρέπει να ξεχαρίσουμε πως δεν υπάρχει αυτοματισμός ή ε, διακριτικά μέτρα εις βάρος των τρίτων αυτών χωρών και Ελπίζουμε βεβαίω να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα στις ε, διεθνείς μας ε, σχέσεις. Ευχαρίστω να επανέλθω και να σας ενημερώσω περαιτέρω για την κατάσταση στο Συμβούλιο καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις του κειμένου αυτού. Είτε μιλάμε για τις τεχνικές λεπτομέρειες είτε ζητήματα πιο πολιτικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Συγητής, ο κύριος Διαθεμέρα. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να πω πως ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την προθυμία τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου για την ε, διαβίβαση αυτού του φακέλου. Ε, επανειλημμένα υπήρχαν συναντήσεις με το Συμβούλιο και μία επίσης με τον κύριο Λεβούς, του εκπρόσωπο της Κομισιόν. Και τον ευχαριστώ θα πρέπει να πούμε πέραν των όσων αναφέρθηκαν ότι έχει αρχίσει να διαγράφεται και η θέση του συγητή. Μιλάμε για την ε, νομική βάση 2007-2 77.2α της συνθήκης και ο βασικός στόχος της πρότασης, πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η βελτίωση της ε, διαχείρισης, ε, τη μετακίνηση υπηκών τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα προβλέπουμε και την ε, παράνομη χρήση των, μάλλον την, την παράτυπη χρήση των ε, θεωρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού αλλά και να προστατεύσουμε και τα άτομα τα οποία χρήζουν ε, διεθνούς προστασίας. Τώρα, πέραν ε, των τεχνικών διευκρινήσεων, η πρόταση προβλέπει την ρήτρα διασφάλισης, την οποία ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα όχι μόνο να επαναλάβω αλλά να τονίσω κάποια ζητήματα που άπτονται της ε, Ρήτρας διασφάλισης που ε, προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την χρησιμοποίησή της αλλά και για την ενεργοποίησή της. Ε, θα ήθελα να τονίσω πως ε, έχουμε και μια άλλη ρήτρα διασφάλισης στη συνθήκη Λισαβόνας, αυτή αφορά στο άσυλο και που καλύπτεται από το άρθρο 78 Αλλά η ρήτρα που θα εξετάσουμε είναι διαφορετική. Είναι συμπληρωματική της πρώτης, αλλά είναι διακριτή. Και κατά την άποψή μου είναι πιο συγκεκριμένη, πιο σαφής, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική σκέψη. Στην ουσία δίνει μικρότερα περιθώρια και κατά άποψή μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διότι είναι πιο σαφής, λιγότερο γενική λοιπόν και πιο σαφής. Αυτό όμως θα συζητηθεί κατά την όλη διαδικασία αυτού του φακέλου. Λοιπόν, συνοψίζοντα, ε, να πω τα εξή, όλη φορά τη διαδικασία. Κοινοποίηση, αξιολόγηση, πριν από την ενημέρωση των ε, ενδιαφερομένων κρατών μελών της υπηρεσίας ασύλου και του Frontex. Αλλά όχι και ή, αλλά ή. ή. Χρειάζεται λοιπόν ε, να ακολουθήσουμε την ε, οδό της ε, επιτροπολογίας ε, αναφέροντας στην Κομισιόν εκτελεστικές ουσίες σύμφωνα με την συνθήκη αλλά λαμβάνοντας υπόψη πως ο εισηγητής και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα αναφέρουν τις προσφυγές που μπορούν να γίνουν Μέσω των τροπολογιών λοιπόν που θα καταθέσω θα πρέπει να οδηγηθούμε στον πολιτικό σύμβασμο στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τεγκούστο. Αυτό θα ήθελα να το εγγυηθώ και για το λόγο αυτό ζητώ την στήριξη των πολιτικών ομάδων. Κατά την άποψή μου, νομίζω πως η ρήτρα και οι τροποποιήσεις απαιτούν κάποια αποτρεπτικά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν και την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον ε, ενδεχόμενων και διαπιστωμένων ε, απατών και καταχρήσεων. Η ρήτρα λοιπόν διασφάλισης ε, θα βοηθήσει στο να διατηρήσουμε την απελευθέρωση της ε, διαδικασίας ε, θεωρήσεων και θα αυξήσει την αξιοπιστία της. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι ακόμα σε ό,τι φορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας, πρόκειται στην ουσία για ένα μέτρο το οποίο αφορά στην αποκατάσταση της υποχρέωσης ε, χωρίς θεωρήσεων σε ένα κράτος το οποίο δεν εφαρμόζει την ε, εξαίρεση και το μέτρο αυτό δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε καμία περίπτωση ε, μονόπλευρα από τα κράτη-μέλη ούτε και στο πλαίσιο της ε, ρήτρα διασφάλισης θα εφαρμόζεται αυτόματα και εδώ θα απαιτείται μια αναλυτική εξέταση η οποία θα λαμβάνει υπόψη την εξωτερική σφαιρική πολιτική, την σφαιρική εξωτερική πολιτική, τονίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν ε, είναι το, ο πυρήνας ε, του ζητήματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως ο ορισμός των θεωρήσεων θα να τροποποιήσουμε τον κανονισμό για να συντονίσουμε τον ε, ορισμό για να συμπεριλάβουμε τους πρόσφυγες και τους απάτητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθιστώντας σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν ε, επηρεάζονται διόλου από τον κανονισμό 539-2001. Επίσης ε, η αναρμόνιση των υποχρεώσεων και η εξαίρεση θεωρήσεων για ορισμένες κατηγορίες που απαριθμούνται στο 4.1 και που μπορώ να συνοψίσω ως εξή. Τα πληρώματα πλοίων, τα πληρώματα αεροσκαφών και τα πληρώματα πλοίων που κινούνται σε διεθνείς ποτάμιες όδους ε, επίσης φυσικά και τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων. Χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη ε, και οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι δεν είναι διακυβερνητικοί. Ε, έτσι κύριε Πρόεδρε νομίζω πως έθιξα το περιεχόμενο της τροποποίησης είναι η ενάτη, τροποποίηση του κανονισμού που μας απασχολεί σήμερα διότι ήδη έχουν υπάρξει οκτώ τροποποίησεις και στην προηγούμενη ήμουν και εγώ πάντα, πάλι συγητής που αφορούσε την Κίνα και την ε, Ταϊβάν. Θα θέλω να πω Κύριε Πρόεδρε, τώρα κάτι για την ορολογία. Για να διατηρηθεί η συνέπεια με τις τελευταίες αποφάσεις που έλαβε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ορολογίας, να υπενθυμίσω την ανάγκη προσαρμογής τους όρους όταν μιλάμε για μετανάστευση παράνομη ή λαθρέα όπως ε, πράξαμε τα τελευταία χρόνια θα ήταν επιθυμητό να αποσυνδέσουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης ε, από τον όρο παράνομη λαθρομετανάστευσης και έτσι να αποφύγουμε την θυματοποίηση των ε, ατόμων που, που βρίσκονται νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε την έκφραση παράτυπη μετανάστευση ή λάθρο μετανάστευση στην, αντί για παράνομη. Παράτυπη λοιπόν και κάτι ακόμα. Τα δίκτυα και οι διακινητές ε, είναι παράνομοι. Όπως και η εργασία μπορεί να είναι παράνομη. Αλλά τα θύματα όχι. Δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι παρανομούν ή είναι παράτυπα ή είναι ε, θύματα λάθρο μετανάστευσης. Ε, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, πάρα πολλές ε, εκθέσεις ε, από πλευράς Κομισιών, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το νομικό αυτό ζήτημα. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μια λύση μέσω μια σύστασης που θα αναφέρεται στην τη σκέψη εν οποία αρμόδιος και υπεύθυνος είναι ο εισηγητής που να την χάνει τη στήριξη του Κοινοβουλίου και χαίρομαι να πω ότι η Επίτροπος ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει στις κοινοβουλικές συνόδους τον όρο παράνομη. Πάντα η κυρία Βάλστρομ χρησιμοποιεί και γι' αυτό την ευχαριστούμε τον όρο παράτυπη ή λαθρέα μετανάστευση. Αυτά και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή κύριο Ντίας Δεμέρα για την παρουσίαση της εκθέσεως. Αυτό το ζήτημα της ορολογίας ε, δεν είναι κάτι το κοινότυπο. Για ε, μια ακόμα φορά το ζήτημα αυτό ε, συζητήθηκε και τονίστηκε στις συζητήσεις που είχαμε και θα πρέπει να επενθυμίζουμε κάθε φορά που καταφεύγουμε σε διαφορετική ορολογία και μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, θα θέλω να πω ότι έχει συμπεριληφθεί στα νομικά κείμενα το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και όχι της παράνομης. Τώρα, η κυρία ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Καταλαβαίνω το... τη λογική της πρότασης. Υπάρχουν όμως αρκετά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, περιγράφουμε την κατάσταση ως κατάσταση ανάγκης. Αλλά μιλάμε ότι θα ληφθούν ε, αποφάσεις σε τρει μήνε. Αυτό σημαίνει πω ε, για τρει μήνε θα μπορούν να μπαίνουν οι άνθρωποι χωρί βίζε μέχρι να αποφασίσουν οι Βρυξέλλε. Αντιφαντικό μου φαίνεται. Καταλαβαίνω πω υπάρχουν δυσκολίε ε, στι διαβουλεύσει κτλ. και, και εντό του Κοινοβουλίου. Και είμαι σίγουρη πω ο κύριο Ντία ε, Δεμέρο θα έχει να μα πει κάποια πράγματα για το ότι δεν θα μπορέσουμε εμείς να συνδιαμορφώσουμε την απόφαση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κάτι το περίεργο εδώ πέρα. Το ότι χρειάζονται τρει μήνες να αποφασίσουμε και μιλάμε για έκτακτη ανάγκη. Δεν κολλάει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Το κριτήριο είναι αύξηση κατά 50% τουλάχιστον. Σε άτομα τα οποία παραμένουν λαθρέα ή έχουν ε, απορριφθεί ε, οι αιτήσει επανεισδοχή κτλ. Αλλά βεβαίω 50% του 10 δεν είναι πολύ, 50% των 10.000 είναι πολύ περισσότερο. Οπότε εξαρτάται από το... το τι είναι αυτό το 50% ποσοστό, τι είναι ως πράγματος. Δεν υπάρχει κάποιο κατόφλι εδώ. Οπότε δεν έχουμε αυτομάτως μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εάν ε, έχουμε αριθμούς που είναι δεκάδες ή εκατοντάδες σε αντίθεση με το να μιλάμε για χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες. Οπότε το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο όριο προξενεί εντύπωση. Και τρίτον, στον κύριο Δεκλόιστερ, είπε ο κύριος Δεκλόιστερ, κάτι το οποίο καλωσορίζω, πως αυτό δεν αφορά συγκεκριμένες χώρες, ήθελε να μας διαβεβαιώσει πως δεν μιλάμε ειδικά για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά μπορείτε να μου υπενθυμίσετε γιατί ε, έλειπα και μισή μήνα και δεν έχω ακόμα επανέλθει. Ποιες άλλες χώρες στην ευρωπαϊκή γειτονιά ε, έχουν απαλλαγή βίζας. Γιατί από όσο ξέρω καμία βόρειο-αφρικανική χώρα δεν έχει. Οπότε, ποιε είναι οι πίθανε χώρες για τι οποίε μιλάμε. Κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν τις έχω έτσι πρόχειρες. Πλην των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Και η κυρία Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ντεκάστερ και να πω πως συμφωνούμε πως απαιτείται η ρήτρα διασφάλισης, αλλά δυστυχώς καλό θα ήταν να ακούσουμε κάτι περισσότερο από την Κομισιόν για το γιατί επελέχθησαν αυτοί οι όροι για την εισαγωγή του αποκλεισμού ενός κράτους από την απαλλαγή θεώρησης. The case will Μιλήσατε για το ότι θα εξετάζονται οι περιπτώσεις μεμονωμένα, αλλά παρόλα αυτά εισάγονται εδώ πέρα συγκεκριμένα κριτήρια και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και ποσοστά. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει ξαφνική αύξηση κατά τουλάχιστον 50% του αριθμού των παρανόμως διαμενών των υπηκόων. Ε, εξαρτάται από το πόσοι είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας και να εμφανίζεται ένας δεύτερος και μετά έχουμε μία αύξηση 50% λέω μιλήτρια, 100% πράγματι. Τουλάχιστον 50%. Είναι λίγο περίεργο λοιπόν αφενός να υπάρχει πρόθεση να εξετάζονται οι περιπτώσεις μεμονωμένα και απ' την άλλη να υπάρχουν κριτήρια τα οποία πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχουν αυτά τα κριτήρια και όχι άλλα. Συμφωνούμε, εντάξει δεν μπορούμε να αλλάξουμε κατά πολύ το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων, αλλά θα θέλαμε κάποια εξήγηση. Ελπίζω πως με τον κύριο Ντίας Δεμέρο θα έχουμε κάποιες συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και ελπίζω μετά να έχουμε μια ευκαιρία να έχουμε κάποιες περισσότερες ιδέες κατόπιν κ. Ντεκέστερ γνωρίζει πως είμαι ευγνώμων σε ολόκληρη την μονάδα του και σε αυτόν προσωπικά για την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας ατόμων στον κανονισμό 539 του 2006 που είναι οι απάτριδες κάτοχοι διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη είναι οι λεγόμενοι Λετονοί και Εστονοί μη πολίτες. Αλλά, Σάρα, για σένα το λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν ε, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βίζα. Και όταν μιλάμε για απάτριδες, για την, ε, από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα έρθουν στα συμβαλόμενα μέρη αυτού του κανονισμού, καλό θα ήταν να υπάρχει και μία αμοιβαιότητα. Δεν ξέρω. Κύριε Ντεκάστερ, ελπίζω να μπορέσετε να θέσετε το ζήτημα αυτό όταν θα μιλήσετε με εκπροσώπους ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Συνολικά λοιπόν υποστηρίζουμε την ιδέα της ρήτρας διασφάλισης, αλλά θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Με συγχωρείτε. Έχουμε και πάλι μείνει πίσω. Και έχουμε άλλο ένα θέμα ακόμα. Έχουμε άλλο ένα ζήτημα. Για το, το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για τα ναρκωτικά. Οπότε παρακαλώ την Κομισιόν να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο όσο να πιο σύντομα για να τελειώσουμε εδώ πέρα, να ακούσουμε και τον εισηγητή και να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα. Ναι, παρακαλώ λοιπόν Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η τρίμηνη αυτή η περίοδος για να ληφθεί απόφαση για να μιλήσουμε για έκτακτη κατάσταση. Βεβαίω, εντάξει, θα το γνωρίζει ούτω ή άλλω η Κομισιόν πριν από την επίσημη ειδοποίηση. Τρει μήνε είναι το μάξιμουμ, αλλά όπω είπα, δεν υπάρχει αυτοματισμός Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη περίοδος για να αξιολογηθεί η κατάσταση. Και το συνδέω αυτό με το δεύτερο σημείο της Βαρόνης Λάτφορτ. Η αύξηση ε, από 5 σε 10 σε ένα μικρό κράτος μέλος των ε, λαθρέων μεταναστών αυτό καλύπτουμε. Δηλαδή λέμε ότι δεν θα υπάρχει ακριβώς αυτοματισμός. Εάν μιλάμε δηλαδή για ένα κράτος μέλος θα πρέπει να δούμε τον γενικό αντίκτυπο στην κατάσταση ολόκληρης ένωσης. Κατόπιν το θέμα της ανατολικής ε, γειτονίας έχουμε ε, διαλόγους με τη Μολδαβία και την Ουκρανία για απελευθέρωση της ε, βίζας και μπορούμε να ξεκινήσουμε βεβαίως τον διάλογο αλλά μέχρι τώρα πάντα υπήρχε η προϋπόθεση του να λειτουργούν ε, σωστά οι συμφωνίες διευκόλυνσης βίζας και επανεισδοχής. Υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες ήδη με τη Γεωργία, για την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν ε, θα υιοθετήσουμε συστάσεις ή διαπραγματευτικές οδηγίες τον Σεπτέμβριο, αλλά θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όλους. Αλλά Κατά κανόνα περνάμε πρώτα από τη διευκόλυνση και τις συμφωνίες επανεισδοχής. Μετά για τους απάτριδες. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς το οποίο ισχύει για, τα, για τους απάτριδες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία δεν καλύπτει από τον κανονισμό. Γι αυτό, αυτό ακριβώς το παραθυράκι προσπαθούμε να κλείσουμε και αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να υπάρχει υποχρέωση βίζας, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να τους εξαιρέσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε με τους συναδέλφους Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Αλλά δεν συμμετέχουν αυτές οι δύο χώρες, καθώς μιλάμε για κεκτημένο Σέγγεν και αφορά το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομος. Ευχαριστώ. Εάν θέλετε να κάνετε μια σύντομη τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για λόγους αυρότητας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την κυρία Λάτφορντ και την κυρία Στινόκα. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά για να βελτιώσουμε το σχέδιο να υπογραμμίσω κάτι που ανέφερε η Κομισιόν. Είναι διατεθειμένη να κάνουμε τις συνεδριάσεις και τις συναντήσεις που θα είναι απαραίτητες για να αριθμίσουμε τα τεχνικά ζητήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της Μησίας διατάξεως. Πρόκειται για το σημείο 14 κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ με την ε, Επιτροπή ΦΑΜ, η κυρία Μύρια Βασιλιάδου, που είναι συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων. Έχουμε την οδηγία του Απριλίου του 2011 για την ε, πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων ε, που εγκρίθηκε και υπάρχει αναφορά σε, βγαίνει αναφορά στην συντονίστρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπών και η κυρία Μίλια Βασιλιάδου ε, διορίστηκε ως συντονίστρια. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και ευχαριστεί ο πρόεδρος τους διερμηνείς που θα μας παραχωρήσουν πέντε επιπλέον λεπτά. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου για να μας κάνει παρουσίαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με ανέχεστε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Δεν είναι και εύκολο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω με το να σας ευχαριστήσω και για τον ενδιαφέρον σας για την ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης και πρόληψης ε, της εμπορίας ανθρωπίνων όντων και για το ότι ενδιαφέρεστε για τις δραστηριότητε μου. Και θα ήθελα να γνωρίσω τον ρόλο σας ε, και την εργασία σας για την δημιουργία του αξιώματος που κατέχω. Και πράγματι καθίσταται έτσι σαφές πως υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει μια διαφορά στη ζωή των θυμάτων. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου πριν από 6 μήνες και Ελπίζω να μην είναι αδύνατο το έργο μου, δηλαδή να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κρατών μελών, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών στον τομέα τη καταπολέμηση της εμπορία. Καμιά φορά μα ξυπνούν οι αριθμοί θα ήθελα να σα υπενθυμίσω λοιπόν πω η εμπορία ανθρώπων είναι σκλαβιά. Οι αριθμοί είναι συνταρακτικοί. Παγκοσμίω μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους σύμφωνα με τον ΟΗΕ. 80% αυτών των θυμάτων είναι γυναίκες. Και βεβαίως μιλάμε για εκτιμήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα αριθμό που μπορεί να φτάνει και τα 27 εκατομμύρια που είναι αυτή τη στιγμή σκλάβοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Τι σημαίνει αυτό, πως πρέπει να δώσουμε βάρος και στην πρόληψη, δίωξη, προστασία των θυμάτων και συνεργασίες. Και σημαίνει επίσης πως εάν δεν υπάρχει έντονη διάσταση του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα θέματα θα αποτύχουμε. Οπότε η πρώτη μου προτεραιότητα και ταυτόχρονα πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε συνέχεια και συνέπεια και μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδοσιακά δε η σώματεμπορία και η εμπορία ανθρωπίνων όντων ήταν ζήτημα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών όπου βασίζομαι και εγώ. Τα τη μελη είπαν πως δεν είναι πλέον ζήτημα μόνο ποινικό, βεβαίως σαφή σημασία έχει ο νόμος, αλλά πρέπει να υπάρχει και πρόληψη στήριξη των θυμάτων, συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και θέλω να τονίσω τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών εδώ πέρα και ε, βεβαίως εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ε, δημιουργήσω ένα χάρτη συγκεκριμένων πολιτικών. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη εικόνα όλων των διαφορετικών υπηρεσιών και το τι κάνουν και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και συλλέγουμε πληροφορίες ε, όσον αφορά αστυνομική συνεργασία, εμπόριο, εργασιακά, ισότητα των φύλων, ε, υγειονομικές πολιτικές και αυτά είναι μόνο η αρχή. Και βεβαίως ε, μέρος όλων αυτών είναι το να περάσουμε το μήνυμα πως θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Και όταν μιλάμε για συνεργασία μιλάμε μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικών οργανώσεων και οποιοδήποτε ε, είναι σε επαφή με τα θύματα. Η νέα οδηγία που ανέφερε ο Πρόεδρος θα έχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία της Ένωσης και θεωρώ πως στέλνει ένα σαφές μήνυμα μη ανοχή τους εγκληματίες και στήριξη στα θύματα. Βεβαίω πάντα το θέμα είναι η εφαρμογή που θα γίνει σε 1,5 χρόνο από τώρα. Και θεωρώ πως ο ρόλος μου είναι Ξέρετε πως υπάρχουν βεβαίως σε αυτές τις επιτροπές ε, οι διαφορές ε, μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπινών δικαιωμάτων και η οδηγία είναι μια εξαιρετική προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και ο ρόλος μου θεωρώ πως είναι να έχουμε συγκεκριμένο διάλογο μεταξύ των υπηρεσιών μας. Οπότε αυτή τη στιγμή συνιστώ μία ομάδα από διάφορες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μέχρι στιγμής 15 γενικές διευθύνσεις από το εμπόριο, επιχειρήσεις, απασχόληση, έρευνα, για να αναφέρω μόνο μερικές. Ε, μόνο στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που αφορούν τα ζητήματα αυτά άμεσα. Δεδομένου τώρα του χρόνου θα αναφέρω μόνο τα ονόματα των πολιτικών. Αλλά βεβαίω ευχαρίστω να δεχτώ ερωτήσει, Τι έχουμε λοιπόν σκιαγραφίσει και είναι οι εξή, χωρίς σειρά προτεραιότητα. Προτάσει αναδιατύπωσης διαδικασιών ασύλου, οδηγίε ε, συνθήκων υποδοχής, ε, ευρωπαϊκή ατζέντα για τα δικαιώματα του παιδιού, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Ευρωπαϊκή εσωτερική και εσωτερική δράση για τη βία εις βάρος των ε, γυναικών, καταπολέμηση των διακρίσεων, το πακέτο των θυμάτων, η άδεια παραμονής για θύματα σωματεμπορίας από το 2004, η οδηγία περί κυρώσεων, η οδηγία περί εποχικών εργαζομένων, ασυνόδευτη, ανήλικη, το εγχειρίδιο Σέγγεν και ο κώδικας συνόρων Σέγγεν. Όλα αυτά μας απασχολούν και βέβαια όσα σχετίζονται με το έργο μου με τους συναδέλφους στην γενική μου διεύθυνση και παραπέρα για να δημιουργήσουμε περισσότερη συνοχή. Επιπλέον υπάρχουν οι υπηρεσίες, οι 7 υπηρεσίες εσωτερικών και δικαιοσύνης, Europol, Eurojust, το Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων, Frontex, Apple και ESO, το ε, Γραφείο Στήριξης Ασύλου στη Μάλτα. Οπότε, για τις 18 Οκτωβρίου την Ευρωπαϊκή ημέρα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων συνεργαζόμαστε με την ε, Πολωνική Προεδρία και την ε, Κομισιόν για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Επίσης εργάζομαι σε ένα άμεσο σχέδιο ανακοίνωσης που ελπίζω να υπάρχει το δεύτερο τρίμηνο του 2012 για μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Ελπίζω να μην καταλήξουμε να έχουμε πάλι μια λίστα διαφορετικών πρωτοβουλειών απλά για να υπάρχει αυτή η λίστα, αλλά να ασχοληθούμε με ζητήματα που είναι άμεσα και πιεστικά. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε τις ε, διαβουλές που είχαν ξεκινήσει πέρσι με την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με αυτή τη στρατηγική κάποιες από τις ιδέες και βεβαίως αυτή τη στιγμή ε, απλά κατεβάζουμε ιδέες ε, θα αφορούν ζητήματα απασχόλησης οι εργασιακές πολιτικές. Έχουν κέρια σημασία το θέμα της εσωτερικής ε, σωματεμπορίας που ανέφερε η Πολωνική Προεδρία. Το θέμα του διαδικτύου για τη στρατολόγηση θυμάτων που είναι ζήτημα τεράστιο. Βεβαίως η αξιολόγηση των ε, εκστρατιών ε, ενημέρωσης λειτουργών. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Πολύ δουλειά γίνεται, αλλά φαίνεται πως ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην πλευρά της ζήτησης. Πολλά από τα μέλη αυτής της Επιτροπής ήρθαν σε επαφή με την Κομισιόν με ερωτήσεις για το ζήτημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλά και εργασιακής εκμετάλλευσης και το θέμα της ζήτησης. Γνωρίζουμε βεβαίως πως η οδηγία μιλάει για υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των εθνικών νομοθεσιών που ποινικοποιούν τη χρήση των υπηρεσιών που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ανθρωπίνων όντων. Η στρατηγική δεν θα είναι συνολική αν δεν δει το θέμα του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πάμε πέρα από τα λόγια. Οπότε μαζί με τους συναδέλφους στη Γενική μου Διεύθυνση προετοιμάζουμε κάποια έγγραφα για να καταλάβουμε περισσότερο το τι σημαίνει το φύλλο όσον αφορά τις πολιτικές καταπολέμησης ε, της εμπορίας ε, ανθρώπων. Και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από το να τα αναφέρουμε απλώς. Επίσης, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν συνέταξε μια πάρα πολύ πολύτιμη έκθεση για την πληρωμένη αυτή στρατηγική που θα καθοδηγήσει νομίζω το έργο μας, ανέφερα κάποια σημεία ήδη και ζητάμε να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων. Επίσης, είχαμε μια συνάντηση με τους εθνικούς εισηγητές, όπως προβλέπει και πάλι η οδηγία, τον περασμένο Ιούλιο, που βεβαίως ε, βρίσκονται εκεί πέρα για να παρακολουθούν μάλλον για να αναφέρουν τα ζητήματα και τις τάσεις της εμπορίας ανθρωπίνων όντων. Η Κομισιόν είναι συμπρόεδρος στις συναντήσεις αυτές και η τελευταία συνάντηση ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τη συζήτηση της εμπορίας ανθρώπων με την Πολωνική Προεδρία. Επίση. υπάρχει πάρα πολύ αλληλεπικάλυψη με το Συμβούλιο, Συμβούλιο Τη Ευρώπης. Υπάρχει μια σχετική σύμβαση εκεί πέρα, υπάρχει ομάδα γκρέπα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν την εφαρμογή της σύμβασης. Τους έχω ήδη συναντήσει και συζητάμε την δυνατότητα του να μειωθεί η αλληλεπικάλυψη. Να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός και συνοχή και συνεργασία όσον αφορά την οδηγία. Όσον αφορά, δεν μπορώ να διαβάσω και όλη μου την παρουσίαση περνά ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά τα δεδομένα της Ένωσης, το πρώτο ερώτημα που μου κάνουν σε κάθε συνάντηση είναι ποιο, πώς έχει η κατάσταση. Και για να είμαι ειλικρινής, απαντάω πως δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε αρκετά στατιστικά στοιχεία. Έχουμε τα δεδομένα του ΟΗΕ, έχουμε ενδεικτικά δεδομένα από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και αυτά. Βεβαίω η ενερμόνιση των δεδομένων είναι κάτι το πολύ σημαντικό η συλλογή δεδομένων από διαφορετικά κράτη-μέλη είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Οπότε, για τα στατιστικά στοιχεία, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία με την Κομισιόν, τη Γενική μας Διεύθυνση και τη Eurostat να συλλέγουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Μιλάμε μόνο για ένα αρχικό στάδιο και ελπίζω η διαδικασία αυτή να συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό και η Κομισιόν ε, διαθέτει 4 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα ΆΙΖΑΚ για την καταπολέμηση σωματεμπορίας και υπάρχει μία στοχευμένη έκκληση ε, που έγινε στις 22 Αυγούστου. Δεν θα πω περισσότερα τώρα γιατί πιέζει ο χρόνος. Να πω κάτι μόνο για τη χρηματοδότηση και τα έργα συνειδητοποιήσαμε στην Κομισιόν ε, ως ε, τμήμα αυτής της χαρτογράφησης πως πάρα πολλή δουλειά γίνεται από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και στα έργα που αφορούν την εμπορία ανθρωπίνων όντων. Οπότε είμαστε στην ε, διαδικασία του να συλλέγουμε στοιχεία από 9 μέχρι στιγμής γενικές διευθύνσεις και όλες οι πληροφορίες είναι αυτή τη στιγμή στο site της Κομισιόν για λόγους γνώσης, συνοχής κτλ. Και βεβαίως μπορείτε εκεί πέρα να δείτε τα διάφορα έργα και το επόμενο ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά. Οπότε αυτή τη στιγμή σκοπεύω εγώ να προχωρήσουμε σε μια επιθεώρηση όλων των α, πρωτοβουλειών που ισχύουν αυτή τη στιγμή και ε, έλαβαν χώρα στο παρελθόν, να δούμε το τι θα γίνει στο μέλλον και πώς θα προχωρήσουμε με στρατηγικό σχεδιασμό. Εάν ξοδεύονται δηλαδή τα χρήματα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν το ξέρουμε και αυτό πρέπει να μάθουμε. Ανέφερα την ιστοσελίδα και όπως σας είπα, αν δεν θα αναφέρω τώρα τη λίστα, υπάρχουν εκεί πέρα όλα αυτά τα έργα. Τέλος, η εξωτερική διάσταση, και θα είμαι πάλι σύντομη, έχουμε το έγγραφο του 2009 που ήταν μια πρώτη απόπειρα να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή στις δραστηριότητες και η Ουγγρική Προεδρία παρουσίασε το Μάιο του 2011 την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού και το τι κάνουν τα κράτη-μέλη στην τομέα της εξωτερικής δράσης. Και εκεί πέρα και πάλι έχουμε γύρω στις 200 σελίδες ένα φύλλο Excel με όλα τα έργα που χρηματοδοτούν σε τα κράτη-μέλη. Και πάλι λοιπόν καλό είναι να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Έχουν κάποιο νόημα. Μήπως να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτές είναι οι ιδέες τις οποίες ερευνούμε. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως η εμπορία ανθρωπίνων όντων υπάρχει σε διάφορες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο με τις σχέσεις της χώρες της ε, Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, των Δυτικών Βαλκανίων, βεβαίως με την Αφρική, στο σχέδιο δράσης για την Αφρική και βεβαίως ε, το θέτουμε στον διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πάνω από 30 χώρες. Θέλω να ολοκληρώσω εδώ πέρα, ελπίζω να σας έδωσα μια σύντομη εικόνα γιατί ο χρόνος πιέζει αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω για τις προθέσεις μου, για το ότι θέλουμε να υπάρχει μια συνοχή και συντονισμός ε, στις πολιτικές αυτές όσον αφορά το εμπόριο ανθρωπίνων όντων και μίλησα για το πώς θα πρέπει να εστιαστούμε σε εταιρικές σχέσεις, σε συνεργασίες, γιατί αλλιώς δεν θα επιτύχουμε. Οπότε αναμένω τη συνεργασία μαζί σας, σε στενή συνεργασία μαζί σας, για τη διάρκεια της εντολής μου στα πάρα πολύ δύσκολα αυτά καθήκοντα που έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου. Σας ευχαριστούμε για την καλή σας πρόθεση και για την ενθουσιώδη παρουσίαση και σας ευχαριστούμε επίσης που συντομεύσατε την παρουσίασή σας διότι ο χρόνος πιέζει. Και είμαι υποχρεωμένος να ανοίξω τη συζήτηση αλλά αλλά έχοντας υπόψη μας ότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς παρακαλώ δύο λεπτά έκαστος και να πω ότι σας ευχόμαστε κυρία Βασιλιάδου καλή επιτυχία στο έργο σας. Λοιπόν, ο λόγος ε, στα μέλη. Η κυρία Χέντε. το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βασιλιάδου. Το έργο σας ε, είναι σημαντικό και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καθόλου τη διάρκεια της θητείας σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα προκαταρκτικά σας σχόλια αν και έχουμε πολύ λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, αλλά ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και ελπίζουμε να συναντηθούμε επανειλημμένα εδώ στο πλαίσιο της Επιτροπής μας για να μας ενημερώνετε. Ε, χαίρομαι που θίξερε το ζήτημα της ε, πρόληψης ε, επανειλημμένα, διότι είναι σημαντικότατο θέμα, διότι η διασυνοριακή εγκληματικότητα αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δουλέψουμε και να καταπολεμήσουμε την ζήτηση. Ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, κυρία Μάγερ έθιξε το ζήτημα που ήταν και η συγγήτρια. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία όλα τα κράτη-μέλη να είναι παρόντα και να λειτουργήσουν στο μήκο κύματο με τους εθνικούς συντονιστέ όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα πρέπει να ασκήσουν πίεση για να υπάρξει επιτέλους καταπολέμηση αυτής της ε, εμπορίας ε, ανθρώπων. Ευχαριστώ. Το λόγο... Δεν πρόσεξα πώς είχε ζητήσει, πώς έχουμε και την κυρία Πάουρα εδώ πέρα, την ε, συμπρόεδρο. Α, δεν έχει εκλεγεί. Απλά αντικαθιστά κάποιον. Τέλος πάντων, συμπροεδρεύει εκπροσωπώντα την Επιτροπή Γυναικών. Οπότε η κυρία Μπάουερ έχει το λόγο. Thank you so much. I'm really sorry that... Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν ε, μπορώ να πω πολλά λόγια λόγω της καθυστερημένης έναρξης ε, της παρουσίασης ε, από την κυρία Βασιλιάδου και να πω ότι εδώ έχουμε την συντονίστρια και αυτό είναι το πρώτο ενδεχόμενο αποτέλεσμα της πρόσφατα υιοθετηθής ε, οδηγίας και της εύχομαι κάθε επιτυχία διότι το έργο της είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση. Επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα μπορούσατε να ασχοληθείτε επίσης με το θέμα της ε, διακίνησης παιδιών ε, Υπάρχουν και, υπάρχει μια άλλη δυνατότητα λοιπόν να σας συναντήσουμε σε άλλο πλαίσιο και να συζητήσουμε την στρατηγική αυτή και πραγματικά έχουμε μεγάλη έρευνα για αυτήν την ε, στρατηγική κυρία Μπότσουγουντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασιλιάδου, καλώς ήρθατε. Εγώ χαίρομαι, χάρηκα για την παρουσίασή σας γεμάτη έτσι, φιλοδοξία και είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης και η κυρία Μπάουερ είπε πως είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να συμβιβάσουμε τους διάφορους ε, τομείς πολιτικής και τα κράτη-μέλη να έχουν τα μέσα να κάνουν την ε, δουλειά τους. Πρέπει λοιπόν να αποτελέσει σημείο σημαντικό και για την Επιτροπή μας γιατί βεβαίως τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πώς ε, θα ε, γίνει αυτός ο συντονισμός και καλό είναι το ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η αντιμετώπιση από ευρωπαϊκής ε, πλευράς. Κάποιες πρακτικές ερωτήσεις. Δεν μιλάμε ακόμα βεβαίως για ευρωπαϊκό δίκτυο ε, ΜΚΟ που ασχολούνται με αυτό το θέμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως δεν είναι η ίδια η κατάσταση και σε όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά το εμπόριο ανθρωπίνων όντων. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχετε κάποιο όραμα από αυτό. Επίση, μιλήσατε για τις τρίτες χώρε και τι γειτονικέ. Ε, χώρες, ε, οπωσδήποτε οι χώρες ε, προέλευσης ή διέλευσης γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό είναι να δώσουμε και εκεί πέρα βάρος και σε συνεργασία με τις χώρες αυτές να φροντίσουμε να υπάρξει μια πολιτική με τις χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία έτσι ώστε εκεί να έχουμε μια καλή προσέγγιση τέλος να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας με τη Europol και τη Eurojust. Το ερώτημά μου είναι εάν έχουν γίνει βήματα για να, να δείτε τι μπορεί να γίνει και εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ντάχη. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία συντονίστρια και να την παροτρύνω για το να συνεχίσει με ιδιαίτερη ένταση το έργο της τώρα για την Επιτροπή μας η οποία έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη του ζητήματος το οποίο εσείς συντονίζετε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική διαπίστωση και θα σας προτείνω κάποια στοιχεία αν θέλετε φυσικά να τα λάβετε υπόψη σας θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην προσεχή συνάντηση. Το ένα αφορά τις ε, διαδρομές. Υπάρχουν έξι οδοί, ε, ε, χερσαίοι και έξι οδοί διαθαλάσσεις. Θα πρέπει να δούμε, βρούμε λοιπόν την τυπολογία των σχέσεων που υπάρχουν σε οικογενειακό επίπεδο θα μιλήσουμε για τους Νιγηριανούς και για τους Κινέζους θα πρέπει να μιλήσουμε για την εκμετάλλευση των θυμάτων σε τέσσερα επίπεδα στον εργασιακό χώρο, στον σεξουαλικό, στον ε, ε, την εμπόριο παιδιών και το εμπόριο οργάνων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφθορά των αρχών που είναι ένα ζήτημα δίχως, το οποίο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η διακίνηση ανθρώπων και η εμπορία αυτών. Και επίσης να ρωτήσω πώς λειτουργεί το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Παπαπούλου. I shall speak in my native language. Ε, κυρία Βασιλιάδου, σας για τον διορισμό σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στη δύσκολη εντολή που έχετε ενώπιον σα. Από την παρουσίασή σας που ήταν πολύ ολοκληρωμένη και περιεκτική, ε, έχουν απαντηθεί κάποια ερωτήματα μου. Θα αρκεστώ μόνο σε κάποια επισήμανση. Θεωρώ ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 θα είναι πολύ υποβοηθητική στο έργο σας και ε, στέκομαι σε αυτό που έχετε πει όσον αφορά την ανάγκη για συγκριτικά στοιχεία για την εμπορία και κοινού δείχτες για την εμπορία ανθρώπων. Διαρωτούμε ακριβώς τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να έχουμε επιτέλους συγκριτικά γιατί είναι πολύ σημαντικά στον τρόπο δράσης για αντιμετώπιση της εμπορίας. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις νέες μορφές εμπορίας. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ουγγρική Προεδρία έχει μιλήσει για νέες μορφές εμπορίας όσον αφορά την εκμετάλλευση ατόμων σε εγκληματικές ενέργειες και όσον αφορά την αξιοποίηση τους για να ζητιανεύουν. Ε, ρωτούμε σε ποιο βαθμό το νέο τρίο προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολωνία, Δανία και Κύπρος, θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία και να συνεχίσει για να αντιμετωπίσει ακριβώς τις νέες μορφές εμπορίας. Ευχαριστώ. And Η ε, κυρία Μορβάη, δύο λεπτάκια ακόμα πριν ε, μας απαντήσει η κυρία Βασιλιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πρώτο μου λεπτό θα ήθελα να σας πω μια ιστοριούλα. Στο δεύτερο λεπτό θα βγάλω συμπεράσματα. Η ιστοριούλα είναι η εξή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει στο Παρίσι σε μια μεγάλη λεωφόρο και είδα έκπληκτη 50-60 γυναίκες από την Ασία που ήταν προφανώς πόρνες. Το τσέκαρα εκεί πέρα με τους μαγαζάτορες και μου είπανε ναι πράγματι αυτές οι γυναίκες από την Ασία είναι πόρνες. Αυτή η κατάσταση γίνεται εδώ και δύο χρόνια στο κέντρο του Παρισιού. Τι έκανα λοιπόν, πήγα εγώ απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και δεν έκανα τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να προτείνω σε εσά και στους συναδέλφους σας. Παρατηρούσα το τι γινόταν. Σε 30 λεπτά, μία η ώρα περίπου, εμφανίστηκαν δύο σωματώδεις κύριοι και μοίρασαν πακεταρισμένα γεύματα σε αυτές τις κυρίες. Επειδή είμαι ποινικολόγος ε, και φεμινίστρια, που ασχολούμαι εδώ καιρό με ζητήματα όπως η πορνεία και η σωματεμπορία, είμαι πεπισμένη πως ε, εάν ένας αστυνομικός με πολιτικά έβλεπε αυτό το επεισόδιο θα καταλάβαινε την οργανωμένη φύση ε, και θα μπορούσε να την αποδείξει. Έχω κάποιες προτάσεις με βάση αυτή την ιστοριούλα. Πρώτον, βγείτε από τα γραφεία σας, εσείς και οι συνάδελφοί σας, Πηγαίνετε στο Άμστερνταμ, στα κόκκινα φανάρια, παρατηρήστε τι συμβαίνει, μιλήστε με τις γυναίκες ε, ε, που εκδίδονται, μιλήστε με την αστυνομία, αντιληφθείτε την πραγματικότητα. Δεύτερον, ασκήστε πίεση στα κράτη-μέλη για να αποκτήσουν την πολιτική βούληση να κάνουν κάτι κατά της σωματεμπορίας. Γιατί όλο έγγραφα έχουμε, θέσεις εργασίες, λόγια, λόγια, λόγια και καθόλου δράση και υποφέρουν αυτές οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κυρία Βασιλιάδου. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Θίξατε μία σειρά αποστήματα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω πολύ θίξατε το ζήτημα των νέων μορφής ε, εμπορίας ε, όπως η παράνομη υιοθεσία, η οικιακή σκλαβιά, η δουλεία. Ναι, Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά υφίστανται, αλλά δεν ξέρουμε το εύρος, το μέγεθος, ε, η στρατηγική και μάλλον η ανακοίνωση για τα προσεχή έτη είναι ένα θέμα το οποίο θα λάβει όλα αυτά υπόψη τώρα. Τα δίκτυα των εθνικών εισηγητών θέλουν να εξετάσουν περαιτέρω αυτά τα ζητήματα. Μερικά ξεκίνησαν με την Ουγγρική Προεδρία για τις μορφές εμπορίας. Η Εθνική οι εισηγητές ε, επιθυμούν να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις. Το συζητάει το θέμα και η Πολωνική Προεδρία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ε, δραστηριότητες και επίσης ε, θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση. Υπάρχουν προτάσεις από την Κομισιόν όπου είναι ξεκάθαρο πως ζητούμε από όλους να εξετάσουν αυτές τις νέες μορφές εμπορίας, τις οποίες δεν γνωρίζουν πολλά. Τώρα, για τις διάφορες, ε, τα τομείς πολιτικής, ε, για το συντονισμό τους, ναι, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο εμάς αλλά αφορά το σύνολο της Ευρώπης και των δρασεών της. Αυτό που έχουμε είναι ένα δίκτυο, ε, μια ένα δίκτυο που συνδέει με όλους τους συναδέλφους. Εντάξει, τίποτα δεν, δεν είναι τέλειο, τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά ελπίζουμε να βελτιωθεί περαιτέρω. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΜΚΟ ε, θα το σημείωσα και θα το εξετάσω περαιτέρω. Ως πρώτη αντίδραση να πω ότι δεν γνωρίζω κατά πόσο υπάρχει ένα παρομοιοδίκτυο, ίσως ε, να υπάρχει αν μην το γνωρίζω, αλλά θα μπορούσαν να βρεθούν χρήματα για περαιτέρω ανάπτυξη και χρηματοδότηση. Τώρα, για, τις, τα γραφεία, για τις υπηρεσίε, συναντήσαμε τη Europol και τη Eurojust με τον διευθυντή της Europol και τον πρόεδρο του Eurojust. Εξετάσαμε συγκεκριμένους τομείς για περαιτέρω συνεργασίες και η ιδέα είναι να βρεθούν σαφείς τρόποι προκειμένου να συνεργαστούν οι υπηρεσίες και φυσικά με την ε, βοήθεια της Κομισιόν. Τώρα για την συλλογή δεδομένων θα πω ότι δεν υπάρχει σε συντονισμός ε, σε ό,τι αφορά την συλλογή αυτών των δεδομένων, το να συνεργαστούμε με την Eurostat όπως έχουμε ξεκινήσει και η συλλογή δεδομένων βρίσκεται σε μια πιλωτική φάση. Η Eurostat γι' ε, αυτό υπάρχει για την ε, συλλογή στατιστικών, αλλά χρειάζονται εναρμονισμένες στατιστικές. Και τέλος, ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα επίμαχο το θέμα της ε, πορνείας και των γυναικών που τη χάνουν σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Λάβαμε πάρα πολλές ερωτήσεις από τα αξιότιμα μέλη των δύο επιτροπών για το ζήτημα αυτό. Όπου γνωρίζετε η Κομισιόν δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση ε, της πορνείας, κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν. Πάντως έχει ξεκινήσει η μελέτη και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις ε, της ε, ζήτησης το τομέα της και εκμετάλλευσης και τον συσχετισμό με την βία, με τον καταναγκασμό κλπ. Και τα κράτη-μέλη φυσικά θα... Με τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω πάει σε αυτές τις ε, περιοχές, σε αυτούς τους χώρους που αναφέρατε. Θα επανέλθω, θα επιστρέψω, αλλά φυσικά και καταγράφω τα όσα είπατε Προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συνεργασία και θα επανέλθω στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλιάδου και σας εύχομαστε καλή επιτυχία.